Ε, φορτωμένο το πρόγραμμα και θα πρέπει να τηρήσουμε τους χρόνους ε, γιατί ακολουθεί και συνεδρίαση του Συλλογικού Οργάνου των Επιτρόπων. Γι' αυτό δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Θα ήθελα και πάλι λοιπόν να, να σας ευχαριστήσω για την πειθαρχία που δείχνετε. Κυρίες και κύριοι, είπατε εκπρόσωπε, αγαπητοί υπουργοί, υφυπουργοί, αξιότιμοι καλεσμένη, διακεκριμένη καλεσμένοι, Κυρίε και κύριοι. Νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή που σας υποδέχομαι εδώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ μέρους του Πρόεδρου Ταγιάννη που δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα και να κηρύξω τα εγγένεια της, ε, του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου κατά της θανατικής ποινής. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που οργανώνουμε αυτό το συνέδριο, το συνδιοργανώνουμε μάλλον με το Βέλγιο, το Βασίλειο του Βελγίου και μάλιστα ε, το διοργανώνουμε στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το γνωστό ημικύκλιο. Θα ήθελα να απευθύνω θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό όχι μόνο στους υπουργούς ε, υψηλού, υψηλά ιστάμενους, ε, πρέσβεις ε, και πολλούς ε, διακεκριμένους εκπροσώπους από τις χώρες που είναι υπέρμαχοι αλλά και από τις χώρες που είναι πολέμοι της, της κατάργησης θανατικής ποινής. Επίσης, ευχαριστώ θερμά και την οργάνωση μαζί κατά της θανατικής ποινής που μας βοήθησε στην συνδιοργάνωση αυτής της πολύ επίκαιρης και βαρισίμαντης διάσκεψης. Ήρθαμε εδώ λοιπόν για να συζητήσουμε, αλλά όχι για να έχουμε μεροληπτικό, μεροληπτικές ομιλίες. Ήρθαμε εδώ για να ανταλλάξουμε απόψεις, για να αντιληφθούμε άνεση τις και τις επιφυλάξεις του άλλου και να εξηγήσουμε τα θεμέλια των ε, ηθικών μας πεπιθήσεων. Και φυσικά όλοι πιστεύουμε στις αξίες μας και θέλουμε να εξακριβώσουμε την αλήθεια των ε, επιχειρημάτων μας και την αξία των πεπιθήσεων μας. Ε, φυσικά πολλά επιχειρήματα θα παρουσιαστούν γλαφυρά και εύγλωτα ε, κατά της θανατικής ποινής στη συζήτηση τις επόμενες μέρες. Η θανατική ποινή δεν είναι αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο κατά του εγκλήματος, αλλά οδηγεί σε μία αντιστρέψιμη και ανήκει στο βλάβη σε περίπτωση δικαστικής πλάνης. Και μάλιστα η εφαρμογή της θανατικής ποινής είναι αυθαίρετη ε, διακριτική και χρησιμοποιείται μερικές φορές ως πολιτικό όπλο εις βάρος των πολιτικών αντιπάλων. Αυτό είναι τραγικό, αλλά ισχύει. Οπότε το μήνυμά μου προς όλους σας είναι ότι είμαστε μαζί σε όλη αυτή την προσπάθεια, σε όλο αυτόν τον αγώνα, γιατί το σημείο αφετηρίας μας είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ένα οικουμενικό αγαθό α, της ανθρωπότητας, κοινό αγαθό όλων των πολιτισμών, των παραδόσεων και των θρησκειών. Ε, δεν θα πρέπει λοιπόν να, πλήττουμε αυτή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που και να ε, αντιδράσουμε, να μην δώσουμε στον πειρασμό ότι ε, αυτή, αυτό το πρόγραμμα ε, είναι μόνο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και μάλιστα το 1993 το πρωτόκολλο υπαριθμών 6 του, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί ίσως να ήταν το πρώτο δεσμευτικό νομικά όργανο που ε, σε καιρούς ειρήνης ε, ε, κατήργησε τη θανατική ποινή και μάλιστα υιοθετήθηκε από 46 χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πάντως η θέση μας για το θέμα αυτό καθορίζεται όχι μόνο από το γεγονός ότι είμαστε κατά κάποιου θέματος, αλλά είμαστε υπέρ και κάποιων άλλων. Είμαστε κατά της θανατικής ποινής, γιατί είμαστε υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε κάθε περίσταση. Και Πιστεύουμε ακράδαντα ε, ότι αυτή η υποχρέωσή μα απορρέει από την έννοια τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια και περιχαρακώνεται και κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κυρίω στο άρθρο 3, που διακηρύσει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στη ζωή. Η κατάργηση τη θανατική ποινή ε, είναι πολύ χρόνο αγώνα και έχουμε πολλέ προκλήσει και ενώπιον μα. Να σα υπενθυμίσω ότι το 1991, ε, το έτος που το 1981 μάλλον, το έτος που επίσημα καταργήθηκε η ποινή στη Γαλλία, τότε η πατρίδα μου, η κομμουνιστική τότε Τσεχοσλοβακία, έκανε την τελευταία της ε, εκτέλεση θανατικής ποινή. το 1989. Μεταξύ του 1945 και του 1990 πάνω από 1.200 άνθρωποι εκτελέστηκαν. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ήπειρος ε, δεν είναι ακόμη απαλλαγμένη από τη θανατική ποινή. Ακόμη και σήμερα στη Λευκορωσία εξακολουθεί να ισχύει η θανατική ποινή και να γίνονται εκτελέσεις. Και μάλιστα η Εθνοσυνέλευση το Σεπτέμβριο του 2018, 121 χώρες ψήφισαν υπέρ του δικαιοστασίου, του παγκόσμιου δικαιοστασίου κατά της θανατικής ποινής, επιβεβαιώντας αυτή την παγκόσμια τάση για την κατάργησή της. Και το 2017 μόνο τέσσερις χώρες ε, δηλαδή ε, ε, εφάρμοσα το 84% των εκτελέσεων. Βέβαια δεν είναι μονόδρομος αυτή η προσπάθεια και δεν θα πρέπει να το λαμβάνουμε ως δεδομένο και παρά τις επιτυχίες που είχαμε στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική, σε πολλές χώρες ακόμη υπάρχει ο πειρασμός για την διακοπή του δικαιοστασίου ή την εξέταση θανατικής ποινής ως τμήμα της λύσης στην ποινική δικαιοσύνη. Θα πρέπει λοιπόν να αντισταθούμε σε αυτέ τι εκκλήσει να επαναφέρουμε τη θανατική πίνη και στην Ευρώπη. Και στην πατρίδα μου χαιρετίζω τι προσπάθειε του Παγκόσμιου Συνεδρίου και πολλών οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών για να συνεχιστεί ο δημόσιο διάλογο με εκδηλώσει και διάφορε οργανώσει υπεράσπιση τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Συνεχίζουμε λοιπόν την προσπάθεια και στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, πλήρη εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θανατική ποινή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε υιοθετήσει πολλά σημαντικά ψηφίσματα για, την καθολική, για το καθολικό μορατόριο, το καθολικό δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή. Μερικές φορές ε, ήταν πιο περιπτωσιολογικά για συγκεκριμένες υποθέσεις ή χώρες. Είμαστε, επαναλαμβάνω, κατά της θανατικής ποινής σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίσταση. Γι' αυτό το διατρανώνουμε κάθε χρόνο στην ετήσια μας έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο. Και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε τη δέσμευσή μας. Όχι μόνο σε δικαστικές ατιμιγορίες ή σε επικείμενες δικαστικές αποφάσεις. Θέλουμε δικαστικές, ε, δικονομικές εγγύησεις, μειώσεις ε, ποινής ή ε, μετατροπή ποινής, λαμβάνοντας υπόψη τη θέματα ψυχικής υγείας ή ε, την, τα εγκλήματα ανηλίκων. Και ελπίζουμε αυτό το έβδομο συνέδριο να μας δώσει την ευκαιρία να διατρανώσουμε και πάλι ε, την πεποίθησή μας, να ενισχύσουμε την πυγμή μας και την αποφασιστικότητά μας και να σκεφτούμε νέες στρατηγικές, ενδεχομένως και την, την ε, επαφή μας με επιχειρήσεις, με τον ιδιωτικό τομέα και συζητήσεις για μαζί τους. Σας εύχομαι καλή επιτυχία τις επόμενες μέρες και πολλές καρποφόρες συζητήσεις για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Γιατί πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι από τα πιο επίκαιρα, που όχι μόνο θα πρέπει να είναι αντικείμενο συζήτηση, αλλά τα αποτελέσματα αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να εφαρμοστούν παγκοσμίω. Και σα εγγυώμαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξακολουθήσει να είναι πρωτοπόρο σε αυτή τη διαδικασία. Σα ευχαριστώ. Well, and it is my great pleasure. Και με μεγάλη χαρά καλώ την ύπατη εκπρόσωπο, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φεντερίκα Μογκερίνη, να πάρει τον λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε εδώ σήμερα στην αίθουσα Ελομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του οποίου ο ρόλος αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι ζωτική σημασία ε, την εργασία που από κοινού επιτελούμε για να επιτύχουμε την κατάργηση. Και ευχαριστώ και την, ε, τις βελγικές κυβερνήσεις, ε, τους συναδέλφους εδώ στην πρώτη σειρά και όλους εσάς που μέρα και νύχτα εργάζεστε ακάματα για να διαφυλάξετε το πιο πολύτιμο αγαθό που διαθέτει το κάθε ανθρώπινο τη ζωή του. Είναι τιμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση που φιλοξενούμε το Παγκόσμιο Συνέδριο κατά τη θανατική ποινή. Εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε περήφανοι που είμαστε ο μεγαλύτερος χώρος όπου δεν εφαρμόζεται η θανατική ποινή. Η ένωσή μας είναι ένωση αξιών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε να πούμε ποιες είναι αυτές οι ευρωπαϊκές και πανανθρώπινες αξίες. Πρώτα απ' όλα είναι λοιπόν η αξία τη ανθρώπινης ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι σε αυτή την αίθουσα συμμεριζόμεθα λοιπόν την άποψη ότι κάθε ανθρώπινη ζωή μετράει. Δεν έχει σημασία πόσα λάθη μπορεί να κάνει ένα άτομο, πώς ζει τη ζωή του. Πιστεύουμε ότι ένα κράτος ποτέ δεν μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή ενός πολίτη. Η ε, ανταπόκριση, σε, η αντίδραση σε ένα έγκλημα δεν μπορεί να είναι ένα άλλο έγκλημα. Έχουμε ε, ξεπεράσει την ε, αντίληψη του οφθαλμών αντιοφθαλμού. Πιστεύουμε στη δικαιοσύνη και όχι στην εκδίκηση. Πιστεύω ότι το συμμερίζεστε. Πολλοί έχετε επενδύσει πολλά και συνεχίζετε να επενδύετε σε αυτή την προσπάθεια. Για μένα προσωπικά είναι χαρά και τιμή, αλλά και με συγκινεί το γεγονό ότι είμαι εδώ. Γιατί όταν ήμουν Ιταλίδα Υπουργό Εξωτερικών το 2014, έκανα εκστρατεία για να υπάρξει δικαιοστάσιο για την θανατική ποινή και όλοι μαζί χαρήκαμε όταν τα Ηνωμένα Έθνη το τέλος του 2014 ενέκριναν την απόφασή τους κατά τη θανατική ποινή. Εμείς οι Ευρωπαίοι συμφωνούμε ότι η θανατική ποινή είναι ασύμβατη με την ταυτότητά μας. Είναι κατά των θεμελιωδών αξιών και πεπιθήσεων μας. Καμία χώρα που εξακολουθεί να προβλέπει τη θανατική ποινή δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι άλλο όμως μας συγκεντρώνει και μας συνδέει σήμερα εδώ. Όλοι πιστεύουμε ότι πάντα μπορεί να υπάρξει πρόοδος και ότι για να υπάρξουν θετικέ αλλαγέ χρειάζεται και προσωπική και συλλογική δέσμευση. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Η ιστορία του Παγκοσμίου Συνεδρίου κατά τη θανατική ποινή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι υπάρχουν αλλαγέ και είναι δυνατέ. Το πρώτο τέτοιο συνέδριο έγινε σε μια άλλη πρωτεύουσα τη Ένωση. το 2001 στο Στρασβούργο. Έκτοτε, 31 επιπλέον χώρε αποφάσισαν να καταργήσουν την θανατική ποινή. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο αντιλαμβάνονται ότι η ποινή αυτή δεν είναι ποτέ σωστή επιλογή. Όλο και περισσότερε κυβερνήσει αναλαμβάνουν δράση. Και αυτό χάρη σε προσωπικότητες όπως εσείς, ε, την εργασία σας, ε, την αφοσίωσή σας. Και επίσης τη δύναμη που έχουν ε, οι εμπειρίες σα. Το 2018 ο πρόεδρος της Γκάμπια ανακήρυξε μορατόριου. Το Μάιο το Μπουρκίνα Φάσο κατήργησε τη θανατική ποινή. Τον Ιούνιο του 18 τον Μπενίν επίσης ε, διέγραψε την ποινή αυτή από τον ποινικό κώδικα και η Παλαιστινιακή Αρχή επίσης. Και η Καθολική Εκκλησία τον περασμένο Αύγουστο, Αύγουστο δήλωσε ότι χωρίς καμία εξαίρεση είναι απαράδεκτη αυτή η ποινή. Έστειλε λοιπόν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς όλους τους καθολικούς παντού στον κόσμο και τον Οκτώβριο. Η πολιτεία του Ουάσιγκτον έγινε η 20η πολιτεία των ΗΠΑ όπου δεν ισχύει η θανατική ποινή. Και επίσης, να μην ξεχνάμε, ότι το Δεκέμβριο υπήρξε με πολύ ευρία πλειοψηφία υπερψήφιση έκκληση των ΗΠΑ για να υπάρξει μορατόριο. Το 2018 είχαμε λοιπόν σχεδόν κάθε μήνα ενθαρρυντικά νέα. Ας επιχειρήσουμε και το 2019 να τα πάει ακόμη καλύτερα. Να έχουμε ακόμη περισσότερα θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, είναι πολύ υψηλό ο αριθμό ε, των ε, ατόμων που εκτελούνται κάθε χρόνο. Γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε για να σώσουμε περισσότερε ζωέ, στηρίζοντα την κοινωνία των πολιτών, μέσω ψηφισμάτων στα Ηνωμένα Έθνη και μέσω απευθεία δράση και συζήτηση με τι χώρε όπου εξακολουθεί να ισχύει η θανατική ποινή και ιδιαίτερα με εκείνε που ε, εκδίδουν τις περισσότερες στρατηγικές αποφάσεις. Ξέρουμε ότι πολλά άτομα και αρχές δεν συμμερίζονται τις αρχές μας. Αλλά πιστεύω ότι η αξία της ζωής είναι παρανθρώπινη αξία που ισχύει για όλους τους πολιτισμούς και όλες τις θρησκείες. Υπάρχουν ε, πολύ ισχυρά επιχειρήματα κατά της θανατικής ποινής που είναι απόλυτα λογικά. Να αναφέρω δύο. Τα γνωρίζετε. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να τα τονίζουμε τα θέματα αυτά. Πρώτον, η θανατική ποινή δεν είναι αποτρεπτική. Και δεύτερον, είναι μια αντιστρέψιμη όταν ε, έχει θανατωθεί ένα ε, αθώο άτομο. Ας δώσουμε τώρα παραδείγματα. Στον Καναδά. Ο Καναδάς κατήρισε την θανατική ποινή το 1976. Έκτοτε τα ποσοστά ε, δολοφονιών στον Καναδά δεν έχουν αυξηθεί. Άρα η θεωρία ότι είναι αναγκαία θανατική ποινή για να μειωθεί το έγκλημα δεν βασίζεται στα στοιχεία. Δεύτερον, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατο να διορθωθούν λάθη σε κάθε δικαστικό σύστημα. Γενικά στη ζωή είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη. Αλλά θα ακούσετε τις ιστορίες διαφόρων που κινδύνευαν να εκτελεστούν και που τελικά επεδείχθησαν αθώοι. Και τώρα είναι ζώντα παραδείγματα της ανάγκης για κατάργηση. Υπάρχει η ιστορία του Ρέντιστάιτ στο Ιλινόι, που στη δεκαετία του 80 καταδικάστηκε σε θάνατο. Το 2003 ο κυβερνήτης του Ιλινόι μετέτρεψε την ε, ποινή του σε ισόβιο κάθριξη. Και μόνο μετά ο Ρέντι κατάφερε να αποδείξει την αθωότητά του και να απελευθερωθεί. Και ως ελεύθερο άτομο εργάζεται για την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής τον, ε, στην πολιτεία του και το κατάφερε πριν από μερικά χρόνια. Πρέπει να ακούσουμε αυτές τις ιστορίες και μέσω των ε, ιστοριών πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την οτροπία όσων ακόμη στηρίζουν τη θανατική ποινή. Γιατί οι πολιτισμοί και οι νοοτροπίες μπορούν να αλλάξουν. Ε, οι κουλτούρες δηλαδή και οι νοοτροπίες. Ακόμη και αν είναι βαθιά ε, ριζωμένες και φαίνεται αδύνατο να αλλάξουν. Όπως είπατε, α σκεφτούμε πού ήταν η Ευρώπη πριν από μερικές δεκαετίες και πού είμαστε σήμερα. Θα καταλάβετε ότι όσοι σας λένε ότι είναι αδύνατο να αλλάξουν τα πράγματα και ότι κάτι είναι βαθιά ριζωμένο στην κουλτούρα, ξέρετε και η κουλτούρα, οι νοτροπίες αλλάζουν και η νομοθεσία μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει η ε, νοοτροπία και αντίστροφα. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο οι διεθνείς οργανισμοί και κυβερνήσεις. Είναι και για τα άτομα που ακόμη είναι σε πτέρυγες μελοθανάτων. Είναι για όσους επέζησαν και τώρα ε, ενημερώνουν για το πόσο άδικη είναι η θανατική ποινή. Η σημερινή εκδήλωση μα αφορά όλου την κοινωνία των πολιτών και τι οργανώσει, του υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καθημερινά εργάζονται ούτω ώστε να γίνει παρελθόν η θανατική ποινή. Και ξέρετε ότι μπορείτε να βασίζεστε πάντα στη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα θέλουμε να ακουστεί η φωνή μα, η φωνή σα και είμαι πεπισμένη ότι σιγά σιγά, αλλά ελπίζω και αρκετά γρήγορα, θα επιτύχουμε τον κοινό μα στόχο. Έναν κόσμο όπου τα εγκλήματα να αντιμετωπίζονται με δικαιοσύνη και όχι εκδίκηση και όπου η ανθρώπινη ζωή να είναι πραγματικά πανανθρώπινη αξία που να γίνεται παντού σεβαστή και να προστατεύεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Να αξιοποιήσω την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι έχουμε διερμηνία στις 22 γλώσσες της Ένωσης, αλλά επίσης αραβικά και ρωσικά. Με μεγάλη χαρά τώρα καλωσορίζω τον ε, αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Βελγίου, Didier Renders, ο οποίος τώρα θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, ε, κυρίες και κύριοι αρχηγοί των κρατών, κύριοι Πρωθυπουργοί, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να πω ότι είναι προνόμιο για μένα να μπορώ να σας υποδεχτώ στις Βρυξέλλες για το μεγαλύτερο, ε, τη μεγαλύτερη εκδήλωση για την ε, κατάρριξη της θανατικής ποινής παγκοσμίω. Και ε, εκφράζουμε την γνωμοσύνη μας στο Κοινοβούλιο που μας υποδέχεται στο αιμοκύκλιο του για την εκδήλωση αυτή. Το δικαίωμα στη ζωή είναι το πρώτο θεμελιώδες δικαίωμα. Μια ανεφόρον προϋπόθεση χωρίς την οποία η άσκηση άλλων δικαιωμάτων δεν θα είχε κανένα νόημα. Θεωρώ ότι η θανατική ποινή πλήττει ε, στον πυρήνα της την ε, ανθρωπινή αξιοπρέπεια και είναι μια τιμωρία ε, που υποβαθμίζει, είναι απάνθρωπη και είναι και φρικτή. Συμφωνώ λοιπόν με την πεποίθηση του Αλμπέρ Καμί ότι ούτε στην καρδιά των ανθρώπων, ούτε στα ήθη της κοινωνίας υπάρχει θα υπάρχει κάποια ποινή η οποία θα έχει κάποιο νόημα εάν δεν καταργηθεί η θανατική καταδίκη. Γι' αυτό θέλουμε παγκοσμίω να καταργηθεί η θανατική ποινή ω Βέλγιο. Δεν είναι ένα οτοπικό όνειρο, είναι ένα στόχο ο οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια τη δική μα ζωή. Επειδή το Συμβούλιο τη Ευρώπη ενέκρινε τα πρωτόκολλα 6 και 13 για την ε, κατάργηση της θανατικής ε, ποινής, σήμερα στην Ευρώπη έχουμε έναν χώρο όπου η θανατική ποινή είναι σχεδόν εκτός νόμου. Σχεδόν διότι η Λευκορωσία ακόμη δεν έχει ανταποκριθεί στην Εκκλησία μας. Εκφράζω τη θλίψη μου για αυτήν την ε, απουσία και ελπίζω ότι στο, στην 50 επέτειο του Συμβουλίου της Ευρώπης θα προχωρήσουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ήπειρο και θα την καταφέρουμε όπου να μην υπάρχει καμία θανατική ποινή. Επίση, φέτο γιορτάζουμε την 30 επέτειο από την υιοθέτηση του δευτέρου πρωτοκόλου για το Διεθνέ Σύμφωνο για τα Πολιτικά και ε, Αστικά Δικαιώματα. Η έγκριση του πρωτοκόλλου αυτού προβλέπει την οριστική εγκατάλειψη από τα συμβαλόμενα κράτη της θανατικής ποινής ως ε, ποινική καταδίκης. Ε, έκτοτε, η υιοθέτηση του πρωτοκόλλου εμποδίζει την επανεισαγωγή της θανατικής καταδίκης στο ποινικό σύστημα και προσφέρει περισσότερα ε, εχέγγυα από ότι ένα δικαιοστάσιο που θα μπορούσε ανα πάσα στιγμή να ανασταλεί στην ισχύ του. Σήμερα, 86 κράτη έχουν εγκρίνει το δεύτερο πρωτόκολλο, δηλαδή πέντε χώρες παραπάνω σε σχέση με το προηγούμενο Παγκόσμιο Συνέδριο το 2016. Είναι ενθαρρυντικό αυτό, όμως δεν είναι και αρκετό. Δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη πολλές χώρες παγκοσμίω που έχουν καταργήσει την ε, θανατική ποινή ή δεν την ε, εφαρμόζουν καν. Ω μέλο τη ομάδα φίλων ε, του Δευτέρου Πρωτοκόλου, το Βέλγιο καλεί τι χώρε που ε, δεν έχουν λάβει μέτρα για τη θανατική καταδίκη να εγκρίνουν το Δεύτερο Πρωτόκολλο όσο δυνατόν συντομότερα. Διαπιστώνω άλλωστε ότι μεταξύ τη τεράστια ομάδα των χωρών που δεν εφαρμόζουν τη θανατική ποινή υπάρχει τεράστια ε, ποικιλία. Ε, δικαστικών συστημάτων, νομικών συστημάτων, ε, νοοτροπιών, θρησκευτικών δογμάτων ε, και προελεύσεων. Είναι κρίμα μια μικρή ομάδα χωρών να συνεχίζει να εφαρμόζει ακόμα τη θανατική ποινή. Και είναι σημαντικό να ξεκινήσει διάλογο με τι χώρε αυτέ, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε το στόχο μα, τον απότερο στόχο μα, που είναι η, παγκο... η εξάλληψη τη θανατική ποινή παγκοσμίω. Θέλουμε να οργανωθεί μια συζήτηση εντελώ ελεύθερη και ανοιχτόμυαλη και για τη θανατική ποινή και για κάποια συσχετιζόμενα θέματα. Παρελκόμενα. Χθε στη Γενέβη συμμετείχα σε ένα πάνελ υψηλού επίπεδου για το θέμα τη θανατική ποινή, το οποίο ασχολήθηκε με θέματα δικαίου ε, ω προ την μη διακριτική μεταχείριση και την ισότητα. Πράγματι, η θανατική ποινή εφαρμόζεται πολλές φορές με τρόπο ε, που κάνει διακρίσεις μεταξύ των πολιτών, των πλέον φτωχών, των πλέον ευπαθών από οικονομικής άποψης. Αυτοί πλήττονται δυσανάλογα. Άλλες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ξένοι, οι αλλοδαποί, οι, οι αλλοεθνείς, οι, αλλοδα... οι, οι σεξουαλικές μειονότητες, οι γυναίκες, ε, πολλές φορές ε, ε, αναγκάζονται να υποστούν δυσανάλογες συνέπειες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σκοπιά των θυμάτων υπό την ευρεία έννοια τους. Τα δεδομένα που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας μας αφήνουν να υποθέτουμε ότι η θανατική ποινή προξενεί περισσότερα θύματα και μπορεί να επηρεάσει ολόκληρες κοινότητες για πολλές γενιές στο μέλλον. Το Βέλγιο ανησυχεί ιδιαιτέρως ε, με το τι συμβαίνει με τα θύματα τα ε, μη ε, φανερά αυτά που δεν έρχονται στην επιφάνεια της επικαιρότητα. Τα παιδιά ιδίω. Τα παιδιά των οποίων έχουν θανατωθεί οι γονεί. Τα οποία αναγκάζονται να υποστούν μια διπλή τιμωρία, αλλά θα έπρεπε να βρίσκονται στο κέντρο τη προσοχή μα. Ε, χρειάζονται βεβαίω περισσότερε επιστημονικέ μελέτε και δεδομένα για να έχουμε μια συνολική εικόνα για τον αντίκτυπο τη εφαρμογή τη θανατική ποινή και το πώ αυτή εμποδίζει το να ε, ασκήσει κανεί ένα μεγάλο φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα έπρεπε να έχει. Χαίρομαι που το Παγκόσμιο Συνέδριο θα ασχοληθεί με πολλά από αυτά τα σημεία και ευράτω με τις ευκαιρίες για να επανεπιβεβαιώσω την ε, διάθεση και την επιθυμία του Βελγίου να αγωνιστεί κατά της θανατικής ποινή και να επιδιώξει την παγκόσμια κατάργησή της και εξάλληψή της. Εύχομαι σε όλους τους συμμετέχοντες να είναι πολύ ευχάριστο το συνεδριό σας με πρόσφορες και επικοδομητικές συζητήσεις και διάλογο και ελπίζω ότι με τις ανταλλαγές απόψε μεταξύ χωρών που εφαρμόζουν ή δεν εφαρμόζουν την θανατική ποινή να μπορέσετε να πετύχετε πρόοδο στην εξέταση του όλου θέματος, ώστε να περιοριστεί ε, κι άλλο ο αντίκτυπος ε, και η παρουσία της θενατικής ποινή ε, σε διάφορα νομικά συστήματα, ώστε να καταφέρουμε κάποτε στο μέλλον έστω την πλήρη κατάργησή της, που είναι ο απότερος στόχος μας. Σας ευχαριστώ και πάλι, σας εύχομαι μια πρόσφορη συζήτηση και εύχομαι να σας δω όλους στην τελετή λήξης. Uh, Θα ήθελα επ' ευκαιρία να σας εξηγήσω ότι η Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Μογκενίνη, χρειάστηκε να φύγει γιατί σήμερα συνεδριάζει το συλλογικό όργανο των Επιτρόπων. Οπότε έπρεπε να φύγει. Γι' αυτό και είπα ότι ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Θα καλέσω τώρα την ε, το Κρίστα Μόλι, το πρέσβη της Ελβετίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης του Βελγίου, ε, αξιότιμοι υπουργοί, ε, αξιότιμοι υπέρμαχοι της κατάργησης θανατικής ποινής, ε, εκπρόσωποι κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Εκπροσωπώ την κυρία Μπερισβίλ, την κυρία Πασκάλ Μπερισβίλ που δυστυχώς ένα ζήτημα υγεία την εμπόδισε να έρθει σήμερα. Ο Βίκτορ Ουγκό είπε ότι το απαραβίωστο της ανθρώπινης ζωής είναι το ύψιστο δικαίωμα. Και 100 χρόνια μετά την πολύ γνωστή του έκκληση κατά τη θανατική ποινή, η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει στο άρθρο 3 ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία και στην προσωπική του ασφάλεια. Και αν σήμερα ε, βρισκόμαστε εδώ, σε αυτό το συμβολικό χώρο και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη φιλοξενία, ε, είναι με το μοναδικό σκοπό να προασπίσουμε το δικαίωμα στη ζωή για όλους τους ανθρώπους. Η Ελβετία είναι κατηγορηματικά ενάντια στη θανατική ποινή παντού στον κόσμο και σε κάθε περίσταση. Και η... Ε, είμαστε υπέρ τη κατάργηση τη θανατική ποινή και είμαστε υπέρ του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι και προτεραιότητα τη εξωτερική μα πολιτική. Και δεν είμαστε μόνοι και είστε μάρτυρες αυτής της προσπάθειας ε, για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Περίπου 80% των ε, χωρών έχουν συμπεριλάβει στο Σύνταγμά τους το δικαίωμα στη ζωή και αυτή η θετική τάση φαίνεται και από τον αριθμό των χωρών που στη συνέχεια ε, κατέργησαν τη θανατική ποινή μετά την δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών. 103 χώρες έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα και 170 την έχουν καταργήσει de jure ή de facto ή εφαρμόζουν δικαιοστάσιο για πάνω από 10 χρόνια. Και μας χαροποιεί ιδιαίτερο αυτή η θετική τάση. Θα τη στηρίξουμε γιατί είμαστε υπέρμαχοι αυτής της πρόοδου. Και μάλιστα η Διεθνής Γενέβη, η πρωτεύουσα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που βρίσκεται όπως γνωρίζετε στην Ελβετία, μας ε, ενισχύει την πεποίθηση ότι η εσχάτη των ποινών δεν είναι κατάλληλο μέσο ούτε αποτροπής ούτε καταστολής. Επιπλέον υπάρχει ο πραγματικός κίνδυνος εκτέλεσης ενός αθώου. Και μάλιστα στην έκθεση του εικονογράφου Σαπάτ και της ε, δημοσιογράφου Βίρμα στη Νέα Υόρκη το 2017 είδαμε κάποιους πολύ, ε, κάποιες εικόνες, κάποιους πίνακες που μας ε, συγκλώνησαν και μας στεναχώρησαν. Ο κύριος Ντούνε Ολατουσάνη, τον οποίο συναντήσαμε στο έκτο συνέδριο, πέρασε 27 χρόνια της ζωής του περιμένοντας την απελευθέρωσή του για, μια, για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, ενώ είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Οπότε η θανατική ποινή με την αναμονή που προηγείται της εκτέλεση και με τα χρόνια που περνά κανεί στην απομόνωση, που είναι πραγματικά ψυχολογικό μαρτύριο που υφίσταται ο κατάδικο και η κοίη του, είναι απαράδεκτα. Και μάλιστα στο 7ο αυτό Παγκόσμιο Συνέδριο η Ελβετία καλεί όλε τι χώρε να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να ευαισθητοποιήσουν το, τους πολίτες τους ε, υπέρ της κατάργησης θανατικής ποινής και κυρίως την νεολαία τους. Γιατί όλοι όσοι είμαστε υπέρμαχοι της κατάργησης και όλοι όσοι δραστηριοποιούμαστε εντός και εκτός αυτής της αίθουσας ε, θα πρέπει να προωθήσουμε και να πείσουμε και αυτούς που διστάζουν, που αμφιταλατεύονται. Γιατί πραγματικά αυτή η ποινή σε καμία περίπτωση δεν είναι πράξη δικαιοσύνης, ούτε ε, εξυπηρετεί την αποκατάσταση. Η, η Ελβετία ε, από το 2017 εφαρμόζει το σχέδιο δράση 2017-2019 για την ε, οικουμενική καθολική κατάργηση της ανατικής ποινής. Και έχουμε ε, τρεις στόχους. Πρώτον, οι χώρες που είναι πέρυσι κατάργησης θα, πρέπει να αυξηθούν και μάλιστα η Βουλή της Μαλαισίας να προβεί σε αυτή την κατάργηση είναι πολύ θαρρυντικό παράδειγμα. Δεύτερο στόχο, λιγότερε χώρε να εφαρμόζουν θανατική ποινή και να περιοριστούν οι εκτελέσει. Μάλιστα, πριν από ένα μήνα απελευθερώθηκε η Ασία Μπίμπι, η Πακιστανή που είχε το 2010 καταδικαστεί στο Πακιστάν για βλασφημία. Αυτό είναι θετικό ιονό η απελευθέρωσή τη. Επίση, οι ελάχιστε παγκόσμιε προδιαγραφέ για την θανατική ποινή θα πρέπει να γίνονται καλύτερα σεβαστέ. Τον Ιράν, μάλιστα, ε, μειώνοντα την ε, θανατική ποινή για εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά μείωσε και τον αριθμό των ε, θανατοποινητών. Επίσης, ε, απευθύνουμε συνεχώς εκκλήσεις προς τα κράτη και κάνουμε διπλωματικά διαβήματα και στα πλαίσια της περιοδικής καθολικής εξέτασης των χωρών. Συνεχίζουμε τις εκκλήσεις μας για την ενίσχυση του δικαιώματο στη ζωή και τη εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και αυτό σε συνεργασία με του εταίρου μα και την κοινωνία των πολιτών. Συνεργαζόμαστε, ανταλλάσσουμε γνώμε, εμπειρογνωμοσύνη, γιατί η θανατική ποινή δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα, δήλωνε ο πρώην Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ. Εθνών Μπανκιμούν. Εστερνιζόμαστε αυτή την άποψη. Θα πρέπει να ενωθούμε ώστε να καταργηθεί η θανατική ποινή, ακόμη και εκεί που ισχύει ακόμη. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη να κάνουν αυτό το επιπλέον βήμα και χαιρετίζω τους εκπροσώπους των κρατών σήμερα εδώ, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή και αυτό που μας ενώνει είναι η ανθρώπινη μας αξιοπρέπεια. Θα ήθελα να σας ευχηθώ να αντλήσετε μεγάλη έμπνευση από το τρίμερο αυτό και Θυμίζοντας τους πίνακες του κυρίου Ντούνε Όλα Σάνι, σας διαβεβαιώ ότι η ελβετική κυβέρνηση θα συνεχίσει τη στράτευσή της υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής και σας εύχομαι μια πολύ επικοδομητική και καρποφόρα συζήτηση. Ευχαριστώ. Και τώρα θα πάρει το λόγο ο κύριο Άντουν Χάλβοσεν που είναι υφυπουργό ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τη Νορβηγία. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Το 2016 η Νορβηγία με υπερηφάνεια φιλοξένησε το έκτο παγκόσμιο συνέδριο κατά τη θανατική ποινή, όπου συμμετείχαν πάνω από χίλιοι συμμετέχοντε. Νομίζω ότι είμαστε ακόμη περισσότεροι εδώ σήμερα. Πολλοί συμμετείχατε για να βοηθήσετε να συμβάλλει το Παγκόσμιο Συνέδριο στο Όσλο στην αλλαγή τη πολιτική και των πρακτικών. Από το Όσλο είχαμε θετικέ εξελίξει σε πολλέ χώρε όπως η Γκάμπια, η Μπουρκίνα Φάσο, αλλά και η Μαλαισία. Ε, καταδείξατε τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί αν, υπάρξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση και ισχυρή ηγεσία. Η πρώτη περιφερειακή, το πρώτο Περιφερειακό Αφρικανικό Συνέδριο που έγινε πέρσι στο Αμπιτζάν κατά τη θανατική ποινή πάντα ήταν σημαντικό βήμα Νορβηγία. Με χαρά στήριξε αυτή την εκδήλωση. Το συνέδριο ε, ήταν χώρο επικοδομητικών συζητήσεων και κατέδειξε ότι υπάρχει ισχυρή στράτευση τη νεολαία και τη επόμενη γενιά των αντιπάλων τη θανατική ποινή. Ένα άλλο σημαντικό βήμα ελήφθη τον περασμένο Δεκέμβριο όταν ε, είχαμε ένα ψήφισμα των ΗΠΑ για να υπάρξει μορατόριο κατά τη θανατική ποινή που εγκρίθηκε με ρεκόρ 121 κρατών μέλων ω μέλο του πυρήνα των κρατών που το στήριξαν. Η Νορβηγία ευχαριστεί όλου όσου ε, έλαβαν μέρο και ψήφισαν και είναι αποτέλεσμα τη ε, συνολική τάση κατά τη θανατική ποινή. Όμω υπάρχουν ακόμη πολλέ θανατικέ ποινέ και εκτελέσει σε διάφορε χώρε. Και αυτό μα ανησυχεί. Η θανατική ποινή είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο μία περιοχή, παράδοση, νοοτροπία ή πολιτισμό ή θρησκεία. Κάθε θανατική ποινή, κάθε εκτέλεση είναι μία παράδειγμα τραγωδία. Η Νορβηγία ε, είναι κατά κάθε θανατική ποινή. Αυτό είναι θέμα αρχή για μα. Ωστόσο, κάποτε η θανατική ποινή ήταν ε, βασικό στατικό στοιχείο και του δικού μα ποινικού συστήματο. Τελευταία εκτέλεση έγινε το 1948 από το 1979 η θανατική ποινή έχει καταργηθεί για όλα τα εγκλήματα. Σήμερα η παράγραφος 93 του Νορβηγικού Συντάγματος λέει «Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή, κανείς δεν μπορεί να καταδικαστεί εις θάνατον». Κυρίες και κύριοι, τα κράτη έχουν ε, υποχρέωση να εξασφαλίζουν την ασφάλεια, ευημερία και εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Το σύστημα ποινική δικαιοσύνη πρέπει να διασφαλίσει ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα πρέπει να τιμωρούνται. Αλλά βασική αρχή πρέπει να είναι να του βοηθήσουμε να ε, παρενταχθούν στην κοινωνία. Η θανατική ποινή το καθιστά δύνατο αυτό, γιατί είναι απόλυτη, μη αντιστρέψιμη και μη επανορθώσιμη. Χρειαζόμαστε περισσότερη γνώση και περισσότερη ε, συνειδητοποίηση των σχέσεων μεταξύ της ε, φτώχεια, των διακρίσεων και τη διαφορετική αντιμετώπιση από την ποινική δικαιοσύνη. Η έρευνα δείχνει ότι το, η θανατική ποινή εφαρμόζεται δυσανάλογα κατά μειονοτήτων. Ακόμη και τώρα, στο 2019, άτομα μπορούν να καταδικαστούν θάνατο μόνο και μόνο ε, για ποιον αγαπούν ο, το φίλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η θρησκεία, η εθνότητα, η οικονομική και οικονομική κατάσταση δεν πρέπει να καθορίζουν ποιο καταδικάζεται σε θανατική ποινή. Το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα είναι προκλήσει που όλοι αντιμετωπίζουμε. Χρειαζόμαστε διεθνή συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε. Χρειαζόμαστε αποτροπή, αλλά η θανατική ποινή δεν είναι το τμήμα τη λύση. Η θανατική ποινή δεν οδηγεί σε μείωση τη εγκληματικότητα. Δεν έχουμε στοιχεία ότι έχει αποτρεπτική αξία. Το Παγκόσμιο Συνέδριο πρέπει να συζητήσει αναλυτικέ λύσει. Ευχαριστώ του ε, οικοδεσπότε μα το Βέλγιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και του οργανωτέ. Την οργάνωση μαζί κατά τη ε, θανατική ποινή και τον παγκόσμιο συνασπισμό κατά τη θανατική ε, ποινή. Και ευχαριστώ και του μάρτυρε που έχουμε δώσει, ευχαριστώ που συμμερίζετε τι ε, εμπειρίε σα μαζί μα. Το Παγκόσμιο Συνέδριο είναι ένα χώρο όπου και οι υπέρμαχοι και οι αντίπαλοι τη θανατική ποινή μπορούν να συζητήσουν οικονομικά και όπου τα κράτη, τα ΗΕ ΕΕ και οι περιφερειακέ οργανώσει, κοινωνία των πολιτών και τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα συνεννοούν τι προσπάθειέ του. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τι επόμενε μέρε όσο μπορούμε περισσότερο με βάση το θετικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε στο Όσλο, τη Νέα Υόρκη και φυσικά και στο Αμπιτζάν. Στόχο μα πρέπει να είναι να ανεληφθούν συγκεκριμένα βήματα για να καταργηθεί η θανατική ποινή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Και τώρα θέλω να προσκαλέσω τους επόμενους δύο προσκεκλημένους μας. Πρώτη. Πρώτο πρώτος ο εκτελεστικός διευθυντής ε, του ECPM, ο κύριος Χάζαν, του όλοι κατά της θανατικής ποινής, Ασόμπλε Κοτρέλα Πέντιμορ, και η κυρία Μινάτα Νιακάτα. Τι χαρά, τι χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Τι ευτυχία. Τι ευτυχία να βλέπω τόσα πρόσωπα. Φιλικά πρόσωπα. Πρόσωπα που ε, ε, είναι υπέρ της κατάργησης. Και τι θέληση. Τι θέληση πρέπει να έχετε για να έρχεστε και εσείς, οι εκπρόσωποι των χωρών που δεν έχουν καταργήσει θανατική ποινή, για να μπορείτε να συζητήσετε μαζί μας, να ανταλλάξετε ιδέες. Είναι τιμή. Είναι τιμή για τον οργανισμό μας, τον ECPM, μαζί όλοι κατά τη θενατικής ποινή, να σας υποδέχεται εδώ. Είναι χαρά και τιμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν στην οργάνωση του, ε, του, του σημερινού συνεδρίου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τέλιτσκα, τον αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, που μας έχει υποδεχτεί εδώ σε αυτό το θαυμαστό ημικύκλιο. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μογκερίνη, την είπατε εκπρόσωπο για τις εξωτερικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ευχαριστώ, Ντιτιέ. Ε, ευχαριστώ το Βέλγιο για την υποδοχή του, για την υποστήριξή του. Σας ευχαριστώ, Αουντούν Χάλβορσεν, για την υποστήριξη της Νορβηγίας όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ τον ε, πρεσβευτή της ε, Ελβετίας που όπως είπατε εκπροσωπεί την Ελβετία ως χώρα που προστατεύει πάνω απ' όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ όλες τις χώρες που υποστηρίζουν το συνέδριο και κυρίως την Διεθνή Συμμαχία. Ε, μέλη του Διεθνού Συνασπισμού, του Διεθνού Συμμαχίας, εκπροσωπείτε όλοι σας ό,τι καλύτερο έχουμε στον κόσμο. Αυτόν τον αγώνα για την αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη ζωή. Ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω γιατί δίχως εσάς τους ε, σπόνσορες και υποστηρικτές του συνεδρίου η ομάδα μας, στην οποία θέλω επίσης να πω τη δεν θα μπορούσε να οργανώσει αυτό που σήμερα ζούμε. Χάρη σε εσά, σε όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ, φίλοι μου που είστε υπέρ της κατάργησης, θέλω να απευθυνθώ. Είναι τιμή μου να μπορώ να σας ανακοινώσω ε, επισήμω την παγκόσμια κατάρριξη τη θανατική ποινή και έναν κόσμο που θα έχει απελευθερωθεί πλήρω από τη θενατική καταδίκη. Διότι ό,τι και αν κάνουμε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε λίγα χρόνια θα το πει αυτό, θα ακουστεί αυτή η κουβέντα. Σας βεβαιώνω ότι τώρα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Εάν έχετε αμφιβολίες, Αρκεί να δείτε σήμερα με τι ε, αντίκτυπο, ε, τι επίδραση ασκεί ε, η παρουσία μας σε αυτό το ημικύκλιο του Ευρωκοινοβουλίου. Η αίθουσα είναι κατάμεστη ανθρώπων, πολιτικών ενθυνοδών που λαμβάνουν κέρυες πολιτικές αποφάσεις, βουλευτών, διπλωματών, που θέλουν την κατάργηση, θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα. Εάν έχετε την παραμικρή αμφιβολία, αρκεί να κοιτάξετε τι δρόμο έχουμε διανύσει σήμερα. Ο Βικτόριο Γκο έλεγε στο λεγόμενα, ε, στα λόγια και πράξεις, ότι δεν γίνεται να μιλήσει κανείς για τη θανατική ποινή χωρίς να αναφέρει τον Βικτορικό. Ο 18ο, ο 17ος αιώνας κατήργησε τα βασανιστήρια. Ο 19ος προέβλεπε θα καταργήσει τη το βασανιστήριο. ο 19ος αιώνας κατήργησε τη δουλεία. Έτσι αποδείχτηκε. Ο 20 Ο 20 επικεντρώθηκε στην ισότητα ανδρών γυναικών. Ήρθε λοιπόν η στιγμή. Ο 21ος αιώνα είναι να γίνει αυτός της παγκόσμιας κατάργησης της θανατικής ποινής. Εάν αμφιβάλλετε αρκεί να δείτε τι υποστήριξη έδειξαν τα κράτη στην ε, παγκόσμια συνέλευση του ΟΗΕ όταν ψηφίσαμε για το δικαιοστάσιο. Τρία τέταρτα των κρατών του ΟΗΕ ε, υποστηρίζουν την κατάργηση. Είναι ένας δίκαιος αγώνας ο αγώνας μας λοιπόν. Κάποιοι θα υποστηρίξουν το αντίθετο. Θα επικαλεστούν την εθνική κυριαρχία, την ε, ένομη άσκηση αντιπίνων την ε, δημόσια τάξη που δεν θα είναι ποτέ απολύτως έτοιμη, την ε, απόκριση, την αντίδραση στη βία με βία. Θα ήθελα όμως να απευθυνθώ κατά κύριο λόγο σε εκείνους ακριβώς, σε όσους από εσά δεν είστε πεπισμένοι ακόμη για το πόσο ο αγώνας μας είναι δίκαιος. Θέλω να απευθυνθώ στους πολυάριθμους πρέσβεις εδώ και εκπροσώπους των χωρών που είναι κατά της κατάργησης και που κάνουν το συνέδριο αυτό είναι ένας τόπος συνάντησης μοναδικός στον κόσμο, που μπορούμε να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε ιδέες. Σας προσκαλώ να έρθετε να συζητήσουμε μαζί μας τις επόμενες ημέρες, να ε, επικοινωνήσετε και να μας προσκαλέσετε. Θέλουμε να αναπτύξουμε διάλογο μαζί σας, θέλουμε να προχωρήσουμε στον δρόμο της κατάργησης της θανατικής ποινή. Κάποιοι, λόγου χάρη, έχουν την παράξενη ιδέα ότι δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε στην κατάργηση, διότι οι κοινέ γνώμε στι διάφορε χώρε δεν το θέλουν. Θα αναφέρω τα λόγια του στρατηγού Ντεγκόλ, ο οποίο έλεγε στα απομνημονεύματά του του πολέμου ότι τα πάντα μπορούν κάποια μέρα να συμβούν. Ακόμη και μία ε, απόφαση που έχει να κάνει με την τιμή και την ε, με το φιλότιμο να καταλήξει να είναι μια σωστή πολιτική επένδυση. Αυτήν την πολιτική επένδυση λοιπόν να εκμεταλλευτούμε, την κατάρριξη της θανατικής ποινή. είναι πράξη τιμής και φιλοτίμου. Ποτέ καμία χώρα δεν οπισθοδρόμησε. Αυτή τη στιγμή σπαγιώθηκε στο νόμο η κατάρρευση τη θανατική ποινή. Η κοινή γνώμη ακολουθεί ό,τι και αν γίνει, σε όποια χώρα και αν έγινε αυτό, σε όποια ήπειρο. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην κάνουμε εργαλείο την θανατική ποινή. Δεν είναι αποτρεπτική η θανατική ποινή. Το γνωρίζετε ήδη καλά. Οι μελέτες ε, το δείχνουν. Ε, όπως και η κοινή λογική. Ωστόσο, ε, παραμένει κατά τη διαστολή μία άσκηση, μορφή άσκησης βίας του κράτους εις βάρος των πολιτών του μπορεί να είναι ένα ε, εργαλείο, ένα όπλο για να ασκήσει κανείς καταχρηστικά την εξουσία. Η θανατική ποινή δεν είναι καθόλου πολιτιστική έκφραση, καμιά πολιτιστική έκφραση. Η Ευρώπη, που είναι την γενετήριο δύναμη υπέρ τη κατάργηση, ήταν η καρδιά που χτυπούσε δυνατά, πολλέ φορέ μάλιστα μάτωσε για τη θανατική ποινή. Η Λεμιτόμο είναι γαλλική και ο Πέλεκη ε, αγγλικό. Όμω το κίνημα υπέρ τη κατάργηση ε, ήρθε και από άλλε υπήρου. Η Κίνα σήμερα είναι η πρώτη χώρα εκτέλεση ε, στον κόσμο. Όμω, κατά τη διάρκεια τη δυναστεία Τόγκ, ε, μεταξύ 7ου και 9ου αιώνα, είχε καταργήσει τη θανατική ποινή. Η, Ιαπωνία, που είχε επηρεαστεί από το Κινέζικο οικονομικό σύστημα, είχε καταργήσει τη θανατική ποινή κατά την περίοδο Αιγιάν. Ε, τα πράγματα άλλαξαν όμως δεν μπορούμε να λέμε παρόλα αυτά ότι δεν είναι εφικτό. Η Λατινική Αμερική είναι η πρώτη ήπειρος που έδειξε ευαισθησία για την κατάργηση. Το Μίσιγκαν, ε, η πολιτεία του Μίσιγκαν, από το 1846 την έχει καταργήσει. Θα το δείτε και στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί ε, μετά την ομιλία μου. Μπορέσαμε να αποδείξουμε στο προπαρασκευαστικό συνέδριο του Αμπιτζάν τον περασμένο Απρίλιο ότι η εφαρμογή της θανατικής ποινή στην Αφρικανική Ήπειρο ε, εισήχθη ε, ως επιτοπλίστων από τους διάφορους αποικιοκράτες του παρελθόντος. Η κατάργηση ε, και κάποιες φορές η συγχώρεση, η αμνηστία ε, ήταν οι συνήθεις πρακτικές στην Αφρικανική Ήπειρο. Θέλω να απευθυνθώ και στους ε, πολιτικούς ηθήνοντες των χωρών για, που συμμετέχουν στο δικαιοστάσιο για την εφαρμογή τη θανατική ποινή. Δεν αρκεί αυτό ω λύση. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτήν την κατάσταση. Ένα δικαιοστάσιο, ένα μορατόριο δεν μπορεί παρά να είναι ένα βήμα, ένα στάδιο προ την τελική κατάργηση. Είναι σαν να μένουμε στα μέσα του ποταμού να τον διασχίζουμε και τελικά να καταλήγουμε να μα παρασέχει το ρεύμα. Είναι σαν να συνεχίζουμε να αφήνουμε του μελοθανάτου ε, σε ξεκρέμαστο μπροστά σε μια προοπτική εκτέλεση τη ποινή του. Είναι ψυχολογικό πλέον το βασανιστήριο και για τους καταδικασμένους και για τις οικογένειε τους η δύναμη του δικού σας του συνεδρίου ε, είναι να τα πείτε όλα αυτά, να τα πείτε ξεκάθαρα και πολλά άλλα και να τα προβάλλετε, να προβάλλουμε το κίνημα υπέρ της κατάρκησης γιατί αυτό είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην οποία θέλω να ποτίσω φορό τιμής. Είναι η καρδιά που χτυπάει, που πάλετε, η καρδιά του κινήματος που πάλετε. Εσείς βουλευτές, δικηγόροι, εσείς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εσείς στρατευμένοι υπέρ της κατάργησης. Η καρδιά του αγώνα μας είναι η ενέργεια η δύναμη με την οποία θα προστατεύσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη ζωή παγκοσμίω. Η κατάργηση παγκοσμίω, διότι το κακό ξεκινάει με την αδιαφορία και την παρέτηση. Για κάποιου η ζωή δεν έχει ίσω κανένα νόημα, αλλά για μα. Τίποτε, τίποτε, τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τη ζωή. φίλοι υπέρμαχοι της κατάργησης της θανατικής ποινής. Εξοχότατε καλεσμένοι. Αγαπητοί, φίλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν μπορείτε να διανοηθείτε πόσο χαίρομαι που βλέπω τέτοια θρώα προσέλευση ομίγυρη, γεμάτη ηθήνοντες πολιτικούς, διπλωματικούς, πρέσβεις, προσωπικότητες με επιρροή και με πυγμή να προωθήσουν τον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Είμαστε αποφασισμένοι ο χάρτης που είδαμε του κόσμου σήμερα να γίνει στο μέλλον καταγάλανος, να καταργηθεί παντού η θανατική ποινή. Όλο και περισσότεροι προσχωρούμε στο κίνημα υπέρ της κατάργησης και δίνουμε ραντεβού σε αυτά τα παγκόσμια συνέδρια της οργάνωσής μας μαζί κατά της θανατικής ποινής. Σίγουρα ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε για να φτάσουμε στην κατάργηση είναι μακρύς ακόμη. Στις 20 Φεβρουαρίου, πριν από μία εβδομάδα μόνο, εννέα νέοι άνθρωποι, που μάλιστα δήλωσαν ότι είχαν υποστεί και μαρτύρια για α, εγκλήματα που κατηγορήθηκαν και που δεν είχαν κάνει, εκτελέστηκαν ε, τα χαράματα στην Αίγυπτο. Ενώ α, ακόμη εκκρεμούσε η έφεσή τους ε, και η προσφυγή του στο Δικαστήριο της Αιγύπτου. Βλέπετε ότι ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε είναι μακρύς. Αλλά ελπίζω ότι κάποια στιγμή δεν θα χρειάζεται πια να οργανώνουμε τέτοια συνέδρια. Θα έχουμε τη χαρά να διαλύσουμε και την οργάνωσή μα, το μαζί κατά τη θανατική ποινή. Γιατί χρόνο με το χρόνο και συνέδριο με το συνέδριο, χάρη στη δική σα κινητοποίηση, έχουμε αποτελέσματα. Κάθε χρόνο και μετά από κάθε συνέδριο, οι υπουργοί έρχονται εδώ από διάφορες χώρες για να μας αναγγείλουν την κατάργηση της θανατικής ποινής στη χώρα τους. Και δεν αφιβάλλω ότι ακόμη και φέτος το συνέδριό μας θα είναι ευκαιρία για να ακούσουμε τέτοιες ανακοινώσεις. Και αυτό εξυπηρετεί η οργάνωση αυτή, αυτά τα παγκόσμια συνέδρια, να έρθουν οι χώρες και να διατρανώσουν μπροστά στον κόσμο ολόκληρο, μπροστά στον πλανήτη, ότι η θανατική ποινή που είναι φρικαλέα δεν εφαρμόζεται πια στη χώρα τους και ότι ε, με βάση τις αξίες της κοινωνίας τους δεν επιτρέπεται πια η εκτέλεση κάποιου στο όνομα του λαού, γιατί αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Πάντως ε, οι παρόντες φαντάζομαι όλοι έχουν πιστεί για το δίκαιο αυτό αγώνα. Θα πρέπει τώρα να πείσουμε και τους υπόλοιπους, τους ε, πολέμιους της κατάργησης. Και γι' αυτό τα συνέδριά μας ε, έδειξαν καινοτομίε, δημιουργήσαμε δίκτυα κοινοβουλευτικών υπέρ της κατάργησης, Χρησιμοποίησαμε ακόμη και την, τέχνη ως φορέα ε, του αγώνα μας και φέτος θα δώσουμε έμφαση στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πόρο για την κατάργηση. Μάλιστα, όπως ε, είδαμε κάποια φαρμακευτικά εργαστήρια αρνήθηκαν να δώσουν στην Αμερική σε προϊόντα για για την εκτέλεση χημικά Ακόμη και εταιρείε καλλιτικών συμμετείχαν σε αυτή την ε, εκστρατεία και πολλές άλλες ε, οργανώσεις ιδιωτικέ. Κάθε άνθρωπος, ε, κάθε άντρας, κάθε γυναίκα, κάθε επιχείρηση, κάθε διπλωμάτης, υπουργό, δημοσιογράφος, δικηγόρος μπορεί στο επίπεδό του να δράσει για να προκαλέσει μία αύξηση αυτής της προσπάθεια για την κατάργηση. Ο καθένα βάζει το λιθαράκι του και προσπαθεί να αποτρέψει επέκταση των θανατικών ποινών. Είναι μεγάλος αριθμός των καταδίκων των ανδρών και γυναικών που περιμένουν στο θάλαμο των μελοθανάτων. Θα πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε ε, μια ελπίδα που τους ε, επιτρέπει να επιβιώσουν σε, απέναντι σε αυτό το ρολόι που κυλά και που αναπόδραστα τους οδηγεί στο θάλαμο της εκτέλεσης. Δεν θα πρέπει να καταλήψουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους α, κατάδικους που ε, σκέφτονται ότι θα καπνίσουν το τελευταίο του στιγάρο, το τελευταίο γεύμα, πριν χτυπήσει η λεμιτόμος του θανάτου ε, για μια εκτέλεση που τους έχει επιβληθεί πολύ συχνά και εξαιτία δικαστική πλάνη. Μερικέ φορέ, μάλιστα, αυτοί οι άνθρωποι με την επιμονή του. Ε, είστε εσείς αυτοί που είστε υπέρμαχοι της κατάργησης ε, θα ακούσουμε πολλές μαρτύριες. Πρόκειται για επιζώντες ε, της θανατικής ε, καταδίκης. Είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει στο πετσί τους πόσο επίγει η κατάργηση της θανατικής ποινής. Και πραγματικά το συνέδριό μας είναι ανεξάντλητη πηγή έμπνευση για αυτές τις προσπάθειες. Θα πρέπει να προτείνουμε λοιπόν καινοτόμε λύσεις, ώστε να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να καταλήξουμε στην ολοσχερή και οικουμενική κατάργηση της θανατικής ποινής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η αγιώτης, ο Πάπας Φραγκίσκος, θα μας στείλει ένα σύντομο βίντεο μήνυμα. Saludo a los Θα ήθελα να χαιρετήσω τους οργανωτές και τους συμμετέχοντες σε αυτό το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της θανατικής ποινής που γίνεται στις Βρυξέλλες. Η ανθρώπινη ζωή είναι ένα δώρο που έχουμε λάβει. Το πιο σημαντικό και πρωταρχικό δώρο. Είναι η πηγή όλων των υπόλοιπων αγαθών και δώρων και όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Και ως τέτοιο η ανθρώπινη ζωή αξίζει προστασίας. Ε, και για τον πιστό μάλιστα ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Αλλά και για τους πιστούς και για εκείνους που δεν πιστεύουν, κάθε ζωή είναι ένα αγαθό. Και η αξιοπρέπεια της ζωής θα πρέπει να τύχει προστασίας και σεβασμού χωρίς εξαιρέσεις. Η εσχάτη των ποινών αποτελεί μία μεγάλη παραβίαση και πλήττει αναπανόρθωτα το δικαίωμα στη ζωή που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και αν όντως ισχύει ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες και κοινότητες αντιμετωπίζουν συχνά πολύ σοβαρά εγκλήματα που προσβάλλουν το κοινό αγαθό και την ασφάλεια των ανθρώπων, εξίσου σίγουρο είναι ότι σήμερα έχουμε και άλλα μέσα για να εξηλαιώσουμε την ε, βλάβη που έχει προκληθεί. Και τα σοφρονιστικά συστήματα είναι όλο και πιο αποτελεσματικά για να προστατέψουν την κοινωνία από το κακό που μπορούν να προκαλέσουν ορισμένοι. Εξάλλου, δεν μπορούμε ποτέ να εγκαταλείψουμε την πεποίθηση και να προσφέρουμε στον κατηγορούμενο, ακόμη και στον δράστη, στον αυτοργό των εγκλημάτων, την πιθανότητα, τη δυνατότητα να μεταμελήσει. Και γι' αυτό είναι θετικό ιονός ότι όλο και περισσότερες χώρες προτιμούν τη ζωή και δεν χρησιμοποιούν πια τη θανατική πίνη ή την έχουν εξαλείψει πλήρως από τα δικαιικά τους συστήματα και τα ποινικά τους συστήματα. Η Εκκλησία ήταν ανέκαθεν υπέρ της ζωής και η άποψή της για τη θανατική ποινή έχει οριμάσει και γι' αυτό το λόγο ζήτησε και η κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας να τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την αλλαγή. Για πολύ καιρό θεωρούσαμε τη θανατική ποινή ως κατάλληλη απάντηση στη σοβαρότητα ορισμένων εγκλημάτων και για την προάσπιση του κοινού αγαθού. Παρ' όλα αυτά, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν χάνεται ακόμη και αν έχουν διαπράξει τα φρικαλαιότερα εγκλήματα. Σε κανένα δεν μπορούμε να στερήσουμε τη ζωή και να του στερήσουμε την ευκαιρία να μπορεί να ασπαστεί και πάλι την κοινωνία, την κοινωνία που λάβωσε και που πλήγωσε και που τις προκάλεσε πολλές, πολλά αδεινά. Ο στόχος της κατάργησης ε, της θανατικής ποινής παγκοσμίω ε, αποτελεί ε, μια πολύ γενναία επιβεβαίωση της αρχής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της πεποίθησης ότι ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει το έγκλημα, να αρνηθεί το κακό και να δώσει την, την ευκαιρία σε κάποιον που διέπραξε ένα έγκλημα να μετανοήσει, να ξανασκεφτεί την δράση του και να αλλάξει ενδεχομένω τη ζωή του. Τουλάχιστον να αλλάξει την εσωτερική του κατάσταση. Θα ήθελα να σας συνοδεύσω με τη δέησή μου και να σας εψυχώσω στις εργασίες σας και στις αποφάσεις σας και επίσης να ενθαρρύνω τους ηθήνοντες, τους κυβερνώντες και όλους όσους και όλους όσοι έχουν κάποιες ευθύνες στις χώρες τους να κάνουν τα απαραίτητα βήματα ώστε να καταργηθεί ολοσχερός η θανατική ποινή. Στα χέρια σας βρίσκεται η δυνατότητα να αναγνωρίσετε την αξιοπρέπεια σε κάθε άνθρωπο και να φροντίσετε να μην χαθούν κι άλλες ζωές, αλλά να κερδίσουν αυτές τις ζωές για το κοινό καλό. Σας ευχαριστώ. Uh, ministers, uh, gentlemen. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται έτσι το εναρκτήριο τμήμα της ε, εκδήλωσής μου, μια προσωπική παρατήρηση που θέλω να κάνω. Συχνά προεδρεύω στη συνεδριά της Ολομέλες εδώ στο ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά σήμερα στο χώρο αυτό είχα εντελώς διαφορετική αίσθηση ήταν κάτι ισχυρότερο εδώ από τη συνήθι παρουσία. Υπήρχε κάτι πολύ ισχυρότερο. Και αυτό, μάλιστα, αυτή μου η αίσθηση αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των ομιλιών. Και αυτά που είδαμε στο χάρτη με τα κράτη που έχουν ε, καταργήσει θανατική ποινή, τα εκατοντάδες άτομα που έχουν εκτελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες Βεβαίω ε, επειδή έχουν ε, διαπράξει εγκλήματα. Αλλά υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία δολοφονήθηκαν επειδή ήταν αντιφρονούντε ή εκπρόσωποι κάποιων μειονοτήτων. Αισθάνθηκα ότι η μνήμη τους ήταν παρούσα. Με αυτού ασχοληθήκαμε σε αυτό το δονακτήριο τμήμα. Για άλλη μια φορά εκτιμώ ιδιαίτερα την παρουσία σας Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες μας. Εύχομαι να είναι ενδιαφέρουσες συζητήσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Και είμαι πεπισμένος ότι το έργο μας έχει έννοια εδώ. Και με ενεθάρρυνε και η ενέργεια του ε, προσώπου της οργάνωσης μαζί κατά τη θανάτικη ποινής. Αυτή την ενέργεια χρειαζόμαστε. Βεβαίω χρειαζόμαστε και τους νόμους. Όλα αυτά χρειάζονται σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία και πάλι σε εργασίες. Τώρα παρακαλώ ελάτε για να βγάλουμε όλη μια φωτογραφία μαζί.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 Thank you to the Vice President. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Παύλ Τέλιτσκα, για την αποφασιστική ομιλία του. Ευχαριστούμε που προεδρεύσατε κατά τη διάρκεια της αναρκτήριας ε, εκδήλωσης. Ευχαριστούμε τους υπουργούς, ευχαριστούμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους διακεκριμένους ε, προσκεκλημένους μας. Παρακαλώ καθίστε. Είμαι Μαργαρίτα Σφόρτσα και θα ε, παρουσιάσω το δεύτερο τμήμα της Εκδήλωση. Η συνέντευξη τύπου θα αρχίσει σε μερικά λεπτά, αλλά συνεχίζει το πρόγραμμα Πρώτα απ' όλα, ε, είναι χαρά μου που βλέπω το άτομα εδώ στο κύκλο. Είστε τόσο πολύ σήμερα που χρειάζεται ορισμένοι να παρακολουθούν την εκδήλωση από μια άλλη αίθουσα. Έχουμε πάνω από 1.500 άτομα εδώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας. Λοιπόν, η Βανέσα Πλέης θα πάρει τώρα το λόγο. Είναι δικηγόρος ε, ποινικού δικαίου από την Αμερική, η Βανέσα Πλέης και συγγραφέας. Είναι σημαντική σύγχρονη ποιήτρια. Σήμερα θα μας πει την ιστορία του Κλέιτον Λόκετ. Ο Λόκετ εκτελέστηκε το 2014 στην Οκλαχώμα. Αλλά κάτι δεν πήγε καλά. Μια ε, φοβερή ιστορία και τόσο ανθρώπινη. Μπορείτε να διαβάσετε επίσης και τη μετάφραση των ποιημάτων. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ τη Βανέσα Πλές να έρθει στο βήμα για να μας παρουσιάσει εδώ στο Μικύκλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτήν την εκτέλεση όπου όλα πήγαν στραβά. On April 29, 2014, the Oklahoma Department of Corrections offender Clayton D. Lockett.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 Σας ευχαριστούμε Βανέσα για αυτό το τόσο ε, συγκινητικό πείμα. Όπω είπαμε από την αρχή, ένα ψήφισμα που καλεί σε δικαιοστάσιο για τη θεματική ποινή ε, υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία και με άλλε χώρε στη Γενική Συνέλευση από το 2000, του ΟΗΕ από το 2007. Σήμερα ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο κ. θα μα ε, πει το μήνυμά του για το μορατόριο Και αυτό καλεί σε αναστολή τουλάχιστον αν όχι πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής. I'm pleased to greet this world. Είναι χαρά μου να απευθύνομαι στο Διεθνέ Συνέδριο. Η θανατική ποινή δεν έχει καμία θέση στον 21ο αιώνα. Ε, εκφράζω την, αντίθεσή, την αντίθεσή μου υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Ε, Είμαι περήφανο που η χώρα μου, η χώρα από την οποία προέρχομαι, η Πορτογαλία, κατήργησε από τι πρώτε θανατική ποινή εδώ και 150 χρόνια. Τον περασμένο Δεκέμβριο, το ψήφισμα τη Γενική Συνέλευση που καλεί σε δικαιοστάσιο για την άσκηση τη θανατική ποινή ε, στηρίχθηκε από 121 κράτη. Το μεγαλύτερο αριθμό που έχουμε ποτέ καταγράψει. Καλωσορίζω την πρόοδο, αυτό, πρόοδο αυτή, αλλά δεν φτάνει. Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται παρά την αγριότητά τη και παρά το μύθο ότι είναι αποτρεπτική και παρά το γεγονός ότι πολλοί αθώοι ε, θανατώθηκαν και συνεχίζουν να θανατώνονται. Ο Γενικό Γραμματέα του ΙΕ μαζί με το μεγαλύτερο μέρο των κρατών μελών και τη κοινωνία των πολιτών θα συνεχίσουν να συνηγορούν υπέρ τη παγκόσμια κατάργηση τη θανατική ποινή. Μαζί μπορούμε να την κάνουμε πραγματικότητα αυτή την αλλαγή. Σε τέτοιο πνεύμα σα εύχομαι να έχετε επικοδομητικέ συζητήσει και ε, αναμένω να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε αυτό το κίνημα. 121 countries support. χώρες ε, υπερψήφισαν το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που ζητά δικαιοστάσιο. Εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Σκεφτείτε από πού ξεκινήσαμε. Είναι ένα αποτέλεσμα που δείχνει για μια ακόμη φορά πως η πολιτική θέσμευση κάνει τη διαφορά. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω στο βήμα το πρώην είπα, το για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών πρόεδρο της Επιτροπής ε, των Ηνωμένων Εθνών κατά της θανατικής ποινής, Νάβη Πιλέη. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κυρία Πιλέη. Καλημέρα σε όλους. Είναι τιμή μου που μπορώ να απευθυνθώ ε, στο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά την αναξία δηλαδή, Συνέδριο για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Σήμερα βρίσκομαι εδώ υπό την ιδιότητά μου ως ε, Προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής ε, κατά της θανατικής ποινής, της ICDP. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον κύριο Αντώνιο Ταγιάννη, που οργάνωσε την υποδοχή αυτής της ε, ε, εκδήλωσης σε τόσο εξαιρετικούς χώρους τα μέγαρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να ευχαριστήσω τον είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευρωπαϊκή πολιτική, εξωτερική πολιτική, την κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη, τον κύριο Didier Reinders, ε, υφυπουργό και ε, από την κυβέρνηση του Βελγίου, που ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο και συνδιοργάνωσε το Παγκόσμιο Αυτό Συνέδριο στις Βρυξέλλες, μαζί με την υπεύθυνη με κυβερνητική οργάνωση, τη δική μας, την CPM. από την αρχή είχαμε ε, προσκαλέσει υπουργούς που ακόμα δεν έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή και ήρθαν στην εκδήλωση αυτή Σημειώνω με μεγάλη χαρά ότι το Βέλγιο και άλλε χώρε που συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση, μεταξύ των οποίων η Ελβετία, η Νορβηγία, η Αυστραλία και η Ισπανία, είναι ενεργότατα κρατημέλη ε, τη ομάδα υποστήριξη τη ICDP. Χθες ε, προείδρευσα σε μια ε, παράλληλη εκδήλωση στο Μέγαρο ΕΓΜΟ ε, μια συνεδρίαση μαζί με άλλους επιτρόπους από την ICTP, όπου συζητήσαμε για το πώς τα κράτη καταργούν τη θεματική ποινή και τι διδάγματα μπορούν να αντιληφθούν από τέτοιου είδους εμπειρίες. Ο δρόμος προς την κατάργηση είναι ένα θέμα που συχνά συζητάμε με τους επιτρόπους του ICTP. Από πού να ξεκινήσουμε για το δρόμο προ την κατάργηση. Ο δρόμο προ την κατάργηση δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα. Κάθε, χρο... κάθε χώρα χρειάζεται χρόνο και η SDP πιστεύει ότι η πολιτική ε, ηγεσία και η δράση είναι καθοριστικό παράγοντα για την κατάργηση. Λόγω χάρη, ο πρώην πρόεδρο Ελμπεντότ, που είναι ε, επίτροπο τη SDP και κάθεται εδώ δίπλα μου στην αίθουσα αυτή, ε, έφερε τη χώρα του στο δρόμο τη κατάργηση Και πώς το έκανε. Ανέλαβε πρώτα απ' όλα μια δέσμευση σε διεθνέ επίπεδο εκπροσωπώντα τη χώρα του και προσχώρησε καθώ και κύρωσε το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο στο ICCPR, το οποίο ακολουθήθηκε από την κατάργηση των διατάξεων περιθανατική ποινή από την νομοθεσία τη χώρα του, τη Μογγολία, ώστε η χώρα αυτή να καταργήσει τη θανατική ποινή τελικά πλήρω το 2017. Τώρα όλοι μας έχουμε την ευθύνη βεβαίως να παρακολουθήσουμε πώς πάνε τα πράγματα και δεν θα υπάρξει καμία τάση προς υποτροπή ε, στη Μογγολία και σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι η θενατική ποινή στην κατάργησή της εφαρμόζεται όντως. Χαίρομαι πολύ που ο πρώην Υπουργό ε, τη Γαλλία, Ρομπέρ Μπανταντέρ, ε, και εκείνο επίτροπο τη ICDP, είναι ένα άλλο καλό παράδειγμα ανθρώπου που ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην κατάργηση τη θανατική ποινή στη χώρα του, τη Γαλλία. Υπάρχουν και άλλοι πρωταγωνιστέ που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην κατάργηση στι δικέ του χώρε. Λόγω χάρη στη δική μου τη χώρα, τη Νότια Αφρική. Το συνταγματικό δικαστήριο ε, είχε καταλήξει στην αξιομνημόνευτη απόφαση για, που κατήργησε την θανατική ποινή. Εκεί ο πρόεδρος Μαντέλα είχε προτιμήσει αντί να διοργανωθεί δημοψήφισμα και μετά από τα έντονα συναισθήματα της χώρας όταν ξέφυγε από το Apartheid επιτέλους αποφάσισε να αφήσει την απόφαση στο δικαστικό κλάδο της χώρας ε, το δικαστικό σύστημα, δηλαδή το συνταγματικό δικαστήριο. Είναι ενδιαφέρον ότι και το συνταγματικό δικαστήριο τη Γουατεμάλα έπαιξε ένα τέτοιο ρόλο πολύ πρόσφατα, με μια απόφαση του Νοεμβρίου 2017, που στην πραγματικότητα οδήγησε στην κατάργηση τη θανατική ποινή για συνηθισμένα αδικήματα στη χώρα. Σε χώρε όπω η Ρουάντα, η Αϊτή, η Καμπότζη, το Ανατολικό Τιμόρ. Ε, εμφύλοι πόλεμοι και γενοκτομία που οδήγησαν σε τεράστιες απώλειες ζώων και έχουν σοκάρει όλο τον κόσμο τελικά έφεραν την κατάργηση της θανατικής ποινή, επειδή προσελκύθηκε η διεθνής προσοχή και σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργήθηκαν, ιδρύθηκαν διεθνή δικαστήρια για τα εγκλήματα πολέμου. Το Παγκόσμιο Συνέδριο οργανώθηκε σε μια στιγμή ε, πολύ κέρια. Τη στιγμή που οι προσπάθειες των κρατών μελών, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι προσπάθειες του είπατε προσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέση την οποία ε, είχα για έξι χρόνια, ε, μας έχει επιτρέψει να καταγράφουμε ένα ρεκόρ 121 κρατών μελών που ψηφίζουν υπέρ του ψηφίσματος του ΟΗΕ για το παγκόσμιο δικαιοστάσιο για την κατάργηση τη θανατική ποινή τον περασμένο Δεκέμβριο. Ένα ακόμα βήμα προ την κατάργηση. Είναι να πει κανεί ναι στο μορατόριο. Ταυτόχρονα βλέπουμε τάσει υπέρ τη κατάργηση στην Ήπειρο από την οποία προέρχομαι, την Αφρική. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη με την εξαίρεση τη Λευκορωσία, αλλά και στην Αμερικανική Ήπειρο. Με την εξαίρεση των ΗΠΑ και της περιοχής της ε, Καραϊδικής ε, περιοχές που κατά τα άλλα δεν ε, ε, έχουν τόσες χώρες με θανατική ποινή. Επίσης στην Ασία δισεκατομμύρια ανθρώπων ζουν σε κράτη που ε, τους βαραίνει ως δαμόκλειο πάθη η απειλή της θανατικής ποινής. Υπάρχουν χώρες που διατηρούν τη θανατική ποινή και την εκτελούν. Χιλιάδες άτομα έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στις χώρες αυτές. Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών θεωρούν ότι το να διατηρούν στην νομοθεσία τους τη θανατική ποινή είναι δικαιολογημένο ότι έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα κατά των αδικημάτων που είναι πολύ σοβαρά ή δεν καταλαβαίνουν ότι η αρχή που πρέπει να ακολουθούμε είναι η δικαιοσύνη και όχι η εκδίκηση. Θα ήταν υποκριτικό, όσοι είπατε εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μην αναγνωρίσω και να καταδικάσω τις εκτελέσεις στην Αίγυπτο. 50 μόνο καταδικάστηκαν αυτό το μήνα. Είναι κόλαφος κατά του παγκόσμιο συνεδρίου μας αυτό. Ελπίζω ότι ε, θα συζητήσετε και για αυτό το θέμα. Σε πολλές χώρες, μεταξύ και των χωρών που είναι υπέρ της κατάργησης, Θεωρείται ότι η εθνική κυριαρχία είναι το καθοριστικό στοιχείο για τι αποφάσει σε σχέση με τη θανατική ποινή, όπω αποκαλύπτει η διαρκή συμπερίληψη τη ρήτρα περί εθνική κυριαρχία και όπω αναγκαστικά συμπεριλήφθηκε στο πρόσφατο ψήφισμα για το μορατόριο τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Αυτέ είναι απόπειρε να αφήσει κανεί κατά μέρο την πτυχή τη ανθρωπιά, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ω προ τη θανατική ποινή και να το φέρει όλο αυτό στο επίπεδο μόνο τη ποινική δικαιοσύνη δικαιοσύνη, τη απόδοση ποινική δικαιοσύνη. Είναι πρόκληση για τα κράτη που είναι υπέρ τη κατάργηση να σκεφτούν αν μπορεί να επανεισαχθεί η θανατική ποινή κάποτε. Θα πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε νέε στρατηγικέ, νέε προσεγγίσει, νέα αφηγήματα για να μπορέσουν όσοι εμπλέκονται σε αυτή την προσπάθεια να διατηρήσουν τον αμύωτο ρυθμό ε, υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινή παγκοσμίω. Βάσει της δική μου εμπειρίας και των άλλων εμπειριών, άλλων επιτρόπων του ICDP, πιστεύουμε απόλυτα ότι η κατάργηση της θανατικής ποινή είναι παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στη ζωή. Και είναι και κάτι το αυθαίρετο, διότι πραγματικά περιθωριοποιεί ομάδε του πληθυσμού περισσότερο και υπάρχει πάντοτε και το ενδεχόμενο κάποιος αθώο να εκτελεστεί. Αυτό θα πρέπει να το δούμε ως προς το ότι η θανατική ποινή είναι κάτι που είναι ε, αμετάκλητο. Ε, αυτός είναι και ο λόγος που συμμετείχα στη Διεθνή Επιτροπή κατά της Θανατικής Ποινής. Είχα την τιμή να προεδρεύω από το 2017 και βρέθηκα μεταξύ ε, ανθρώπων εντυπωσιακών μια ομάδα που πραγματικά πιστεύουν βαθιά στον αγώνα υπέρ της κατάργησης και έχουν δείξει πλήρη αφοσίωση και τόλμη στον αγώνα για, την, το σκοπό αυτό στις δικές τους τις χώρες αλλά και διεθνώς. Η Επιτροπή μας διοργανω, ε, ιδρύθηκε βασισμένη στην πεποίθηση ότι η κατάργηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τις κοινέ προσπάθειες κρατών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και διεθνών κυβερνητικών οργανώσεων, δηλαδή κυριολεκτικά όλων ημών μαζί σημερινές συναντήσεις όπως το Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της θανατικής ποινής είναι απαραίτητα ε, για το κίνημά μας. Έτσι ε, δημιουργείται ένα βήμα, μπορούν οι διαφορετικές χώρες να συναντηθούν, να, να εντοπιστούν νέες τάσεις, να συζητηθούν νέες στρατηγικές και νέοι ε, υπεύθυνοι να αρχίσουν να ασχολούνται με το θέμα. Ε, εύχομαι λοιπόν κάθε τύχη από την πλευρά της ICDP στις συζητήσει σας. Ελπίζω να διδαχθούμε εμείς από εσά και το αντίστροφο και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε κυρία Πιλά για τις παρατηρήσεις σας. Όντως υπάρχει μια θετική τάση στην Αφρική υπέρ της κατάργησης και θα το συζητήσουμε σε λίγο με πολλούς καλεσμένους μας. Θα περάσουμε τώρα στα γαλλικά. Θα μιλήσω γαλλικά προς τιμή του επόμενου καλεσμένου μας θα ήθελα να καλωσορίσουμε τον κύριο Ζόρς Ναξέο Γκοφάνκ, ειδικό απεσταλμένο της κυρίας Λουίς Μουσικιβάμπο, που είναι γενική γραμματέας της Διεθνούς Οργάνωσης ε, Γαλλόφωνων Χωρών. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τρία τέταρτα των γαλλόφωνων χωρών μέχρι στιγμής έχουν καταργήσει τη θανατική πίνη. Κυρίες και κύριοι, ε, υπουργοί, εξοχότητες, ε, κυρίες και κύριοι πρεσβευτέ, εξοχότητες προσωπικότητες, ε, διακεκριμένοι καλεσμένοι. Νιώθω τεράστιο προνόμιο και τιμή που θα σας μεταφέρω το μήνυμα της κυρίας Λουίς Μουσικιβάμπο, Γενική Γραμματέα των χωρών, της Διεθνούς Οργάνωσης των Γαλλόφωνων Χωρών, επευκαιρία του 7ου Παγκοσμίου Συνεδρίου κατά της θανατικής ποινής. Ιδού το μήνυμα της κυρίας Μουσικιβάμπο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις ειλικρινέστατες ευχαριστίες μου προς το Βέλγιο που φιλοξενεί αυτή την οργάνωση και στους συνδιοργανωτές αυτού του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου κατά της θανατικής ποινής. Και θα ήθελα να αποδοτήσω φόρο τιμής στις κορυφαίες προσωπικότητες που δέχθηκαν να λάβουν μέρος στο συνέδριο αυτό, προσφέροντας την υποστήριξή τους στον αγώνα για την κατάργηση. Η κοινή μας στράτευση υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής εδράζεται πάνω απ' όλα στην πεποίθησή μας, στην ακράδαντη πεποίθησή μας ότι πρωταρχικό δικαίωμα του ανθρώπου είναι το δικαίωμα στη ζωή, που είναι δικαίωμα αναπαλωτρίωτο. Επίσης, η δράση μας εντάσσεται στη, στο δρόμο της διακήρυξης του Μπαμάκο του Νοεμβρίου του 2000 που υπεθυμίζει τις δεσμεύσεις των χωρών μελών ε, της οργάνωσής μας να σεβαστούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Διεθνή Οργάνωση Γαλλόφωνων Χωρών ε, συντροφεύει αυτέ τι χώρε και τι συμπαρίσταται στι ε, ε, συζητήσει και στι δράσει που γίνονται. Και μάλιστα απευθύνουμε εκκλήσει υπέρ τη κατάργηση τη εσχάτη των ποινών σε συνεργασία με την κοινοβουλευτική διάσκεψη της γαλόφωνίας, καθώς και σε συνεργασία με κάποιες γαλλόφωνες κυβερνήσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Αυτή η όθηση που έχει δημιουργηθεί προς την κατάργηση της θανατικής ποινής έχει μεγάλη απήχηση και στις γαλλόφωνες χώρες. Αυτή τη στιγμή τρία τέταρτα των γαλλόφωνων χωρών έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Και τα τελευταία δέκα χρόνια, οχτώ χώρες μέλη της γαλλοφωνία κατάργησαν τη θανατική ποινή. Και άλλες γαλλόφωνες χώρες αυτή τη στιγμή έχουν δεσμευθεί να καταργήσουν τη θανατική ποινή στο μέλλον. Και ελπίζω ο διάλογος που γίνεται σε αυτό το συνέδριο θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε τα καλύτερα μέσα για να συμπαρασταθούμε στις χώρες που έχουν ακολουθήσει αυτό το δρόμο της κατάργησης της θανατικής ποινής. Επίσης, έχουμε πολύ επικοδομητικές ε, συζητήσεις και σίγουρα τα πορίσματά μας θα είναι πολύ θετικά. Να είστε βέβαιοι ότι και οι γαλλόφωνες χώρες θα λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα του συνεδρίου για να τροφοδοτήσει τις συζητήσεις που θα οργανώσει και τις δράσεις της. Σας εύχομαι πολύ καλές εργασίες. Merci, Monsieur Ευχαριστούμε κύριε Γκοφάνγκ και ευχαριστώ και την οργάνωσή σας, τη Διεθνή Οργάνωση Γαλλόφωνων Χωρών, σε αυτό το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά της Ανατολικής ποινής. Περνάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Φλόριντα είναι από τις πολιτείες που εφαρμόζουν περισσότερες θανατικές ποινές έχουν το, δεύτερο μεγαλύτερο θάλαμο μελοθανάτων ε, των θανατοποιητών που περιμένουν την εκτέλεση. Η κυρία Άραμις, ε, ε, δικηγόρος από την Φλόριντα, δήλωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιδικάσει τέτοια θανατική ποινή. Θα ήθελα να καλωσορίσω και να δώσω το λόγο στην κυρία Άραμις Αγιάλα. It's a great honor to have you with us Μεγάλη μας τιμή, κυρία Αγιάλα. Thank you very much, uh, presidents, ambassadors, diplomats. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και το Βέλγιο που μας φιλοξενεί, προσκύκλοι προσκεκλημένες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου που συμμετέχω στην εκδήλωσή σας και είναι τιμή μου που είμαι εδώ μαζί σας για να προστατεύσουμε τη ζωή και την ανθρωπιά. Τι δικαιοσύνη είναι αυτή όταν όλοι κλείνουμε τα μάτια μας και προσπαθούμε να φανταστούμε πώς είναι δικαιοσύνη. Μπορεί να είναι διαφορετική η δικαιοσύνη όπως τη σκέφτεται ο καθένα, αλλά ο στόχος δικαιοσύνης είναι η ισότητα. Η δικαιοσύνη. Και δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη όταν έχουν προμελετημένη θανάτωση ενός άλλου ανθρώπου που δεν ε, προκαλεί άμεσο κίνδυνο. Η θανατική ποινή είναι η λευκή σημαία τη ε, εγκατάλειψη των προσπαθειών. Όταν επιδιώκουμε θανατική ποινή για όσου δολοφονούν άτομα, λέμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη από την κυβέρνηση. Λέμε ότι δεν μπορούμε να σου δώσουμε το αγαπημένο πρόσωπο πίσω. Οπότε θα πάρουμε μια άλλη ζωή για να αντισταθμίσουμε τη δική σου απώλεια. Παραδεχόμαστε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε δικαιοσύνη στα άτομα τα οποία κινδυνεύουν από τόσο έντονο πόνο. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ε, υπεραντιδρούμε και δεν είμαστε πια ουδέτεροι. Η ουδετερότητα, η αντικειμενικότητα πρέπει να είναι ο βασικός κανόνας δικαιοσύνης. Όταν τη χάνουμε, στην ουσία, εγκαταλείπουμε την ε, λογική σκέψη και υποκύπτουμε στα συναισθήματα. Αποκαλούμε την εκδίκηση δικαιοσύνη, αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη στο θάνατο και η δικαιοσύνη δεν πρέπει να βασίζεται σε συναισθήματα. Όταν τα συναισθήματα εισέρχονται στην ιερή έννοια της δικαιοσύνης, τότε έχουμε αδικία. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι ποτέ η ανθρωπιά. Ως εκλεγμένη εισαγγελέα από τις ΗΠΑ πρέπει να ακολουθήσω το νόμο. Το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας μου απέριψε τις προσπάθειές μου να υπάρξει δικαιοσύνη και να χρησιμοποιήσω τους πόρους όπως επιθυμούσα. Το ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ενδεχόμενο να επιβάλλω θανατική ποινή παρά το ότι είχα πει ότι δεν θα το επιδιώξω. Αλλά ναι μεν θα ακολουθήσω τον νόμο, αλλά πάντα η αλήθεια θα είναι ε, η κατευθύντρια γραμμή μου και θα τονίσω ότι η θανατική ποινή είναι άδικη. Αλλά και όταν ακολουθώ τον νόμο θα συνεχίσω να είμαι άκαμπτη στη θέση μου κατά της θανατικής ποινής. Δεν έχει επικυρωθεί από το νόμο του κράτους μου και ναι, με δεν μου επιτρέπουν να μην αντιμετωπίσω τον δεχόμενο να επιβάλλω θανατική ποινή, αλλά θα συνεχίσω να βασίζομαι στα στοιχεία και ελπίζω κάποια στιγμή στη ζωή μου ο νόμος να συμφωνήσει με τα γεγονότα και όλη την έρευνα που έχουμε για τη θανατική ποινή. Γιατί τα γεγονότα είναι γεγονότα. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι η θανατική ποινή δεν βοηθάει τη δημόσια ασφάλεια. Δεν είναι αποτρεπτική. Για να υπάρχει αποτροπή χρειάζεσαι αυστηρότητα και φυσικά η θανατική ποινή είναι αυστηρία, αλλά η αποτροπή χρειάζεται νομική ασφάλεια και ταχύτητα. Καμία δεν ισχύουν στην περίπτωση θανατική ποινή και πρέπει λοιπόν να εφαρμόζεται ταχύτατα θανατική ποινή. Ξέρουμε ότι οι θανατοποινίτες περιμένουν μέχρι 30 και 40 χρόνια. Οπότε δεν είναι ταχεία η εφαρμογή τη. Επίση, το κόστο που σχετίζεται με την επιβολή της θανατική ποινή είναι τεράστιο. Αλλά δεν το φέρει κανένα από όσου ε, συνεχίζουν με αυτή την αποτυχημένη πολιτική. Το κόστο και το κόστο για την ε, ψυχική υγεία, για αυτού που κάνουν τι εκτελέσει είναι η δουλειά του δηλαδή, αυτά πρέπει να σε ενσυχούν σοβαρά για όλη την ανθρωπότητα είναι ανησυχητικά και το γεγονός ότι όσοι θανατώνουν άλλα όντα υποφέρουν μετά από σύνδρομο τραυματισμού και ψυχική υγείας δεν είναι κάτι που μπορούμε να αγνοούμε. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το γεγονός ότι η θανατική ποινή είναι επίση ε, κάτι που επιβάλλεται με διακριτικό τρόπο και πολλές φορές η διαδικασία έφεσης αποτυγχάνει. Το σύστημα πρέπει να διορθωθεί. Εκπροσωπώ την πολιτεία που είναι μεταξύ των πολιτιών ε, που έχει πολλές φορές, τις περισσότερες φορές από τις περισσότερες άλλες πολιτείες, τελικά αθωώσει άτομα που είχαν καταδικαστεί στην ποινή του θανάτου. Πρέπει να κάνουμε πολύ καλύτερα τη δουλειά μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι δυνατόν να θανατώνουμε άτομα όποια δικαιολογία και αν λέμε. Το να το αποκαλούμε δικαιοσύνη ή να το αιτιολογούμε λέγοντας ότι πάντα έτσι κάναμε, δεν το κάνει σωστό. Είναι μόνο εκδίκηση και δίψα για αίμα που μας κάνει λιγότερο ανθρώπους κάθε φορά που το στηρίζουμε ή που σιωπούμε. Πρέπει να προωθήσουμε την πρόοδο και τη δικαιοσύνη. Κάνοντάς το πρέπει να είμαστε άκαμπτοι και τολμηροί. Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή παρά να αγωνιστούμε από κοινού κατά της θανατικής ποινής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γιάλα για την τόσο θαραλέα τοποθέτησή σας και τον ε, παθιασμένο σας λόγο. Ελπίζουμε και άλλοι και στην Αμερική να σταθούν στο πλευρό σας. Και τώρα πάω κοντά στο πιάνο. Ίσως να ρωτηθείτε γιατί υπάρχει ένα τέτοιο όργανο στο κέντρο του ημικυκλίου του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν έχουμε καμιά κακή πρόθεση. Έχουμε τώρα μαζί μας ένα μεγάλο στάρ του Βελγίου. Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι πήγαν σε συναυλία του και το άλμπουμ του από τότε που κυκλοφόρησε πέρσι είναι best seller. Καλωσορίστε την προσκεκλημένη μας. Thank την Tiff Μπάρο. Ευχαριστούμε Tiff που είσαι μαζί μας. Η Tiff θα τραγουδήσει το τραγούδι La Μπορεί να το ξέρετε. Το έχει συνθέσει ο Μισελ Μπερζέ στην πρώτη του εκτέλεση. Ευχαριστούμε, Τιφ, που είσαι μαζί μας. ξανά το τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. 144 χώρε έχουν καταργήσει βάσει τη νομοθεσία ή στην πράξη την θανατική ποινή. Όμω και πάλι 60% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει κάτω από ένα ε, ποινικό σύστημα, νομικό σύστημα που επιτρέπει τη θανατική ποινή. Εδώ θα ξεκινήσουμε συζήτηση με υπουργού που δέχτηκαν την πρόσκλησή μα, διότι Όπω είπε και ο αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου στην ανακτήρια τελετή, θέλουμε εδώ να ανταλλάξουμε εμπειρίε με όλου. Θα καλέσω λοιπόν στο προσκυνείο την κυρία Τάλατα Αλτοκοράλε, η οποία είναι υπουργό δικαιοσύνη και μεταρρύθμιση των ε, ε, σοφρονιστικών στη Σιλάνκα. Και μετά θέλω να καλέσω και τον κύριο Ζανκλόντ ε, Γκερεσό, ο οποίο είναι υπουργός του Κονγκό, ο κύριος Μεϊξεκό από την Γουινέα και στο πάνελ μας. Θέλουμε επίσης και τον κύριο Μπεσολέ Ρενέ Μπαγκορό, Υπουργό Δικαιοσύνη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προώθηση των Πολιτικών Δικαιωμάτων στην Πουρκίνα Φάσο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αμπομπακάρ Ταμπαντού, ο οποίος είναι Γενικός Εισαγγελέας και Υπουργό δικαιοσύνη στην Γκάμπια και τον Υπουργό Δικαιοσύνη του Μαρόκου, τον κύριο Μοχαμέντ Άουζαρ. Καλώ ήρθατε όλοι σα σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε Υπουργέ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας εδώ στο συνέδριο κατά της θανατικής ποινής. Εάν με επιτρέπετε, θα απευθυνθώ στην κυρία του Κοράλε, την Υπουργό Δικαιοσύνη και Μεταρρύθμιση των Σοφραστικών Ιδρυμάτων στη Σρι Λάνκα. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε στι Βρυξέλλε, Υπουργέ. Διαβάζουμε στον τύπο της Σρι Λάνκας ότι μπορεί και να ξαναρχίσει η επιβολή της θανατικής ποινή μετά από 40 χρόνια συμμετοχή στο μορατόριο. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στη χώρα σας. Πείτε μας. Ladies and gentlemen, dear friends, it gives me great pleasure to thank Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που διοργανώνει αυτή την σημαντική εκδήλωση. Που διοργανώνει αυτό το παγκόσμιο συνέδριο. Σήμερα, καθώς μιλούμε, ε, βλέπουμε ότι το μορατόριο ε, στη Σρι συνεχίζει να ισχύει στην 73η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ψηφίσαμε υπέρ του ψηφίσματος για ένα νέο ε, μορατόριο για τη θανατική ποινή στις 7 Δεκεμβρίου 2018. Πράγμα που είχαμε κάνει και το 2007, 8, 10, 16 επίσης. Μια επιτροπή που διορίστηκε από την κυβέρνηση θα εξετάσει και θα μειώσει τις θανατικές ποινές σε ισόβια ε, κάθερξη, σε ανάλογες ε, περιπτώσεις ή σε μακροχρόνιες φυλακίσεις που θα γίνουν ε, πιο μικρής διάρκειας. Ελπίζουμε ότι οι συνεταίροι μας σε διεθνέ επίπεδο θα καταλάβουν και θα βοηθήσουν τη Σριλάκα να αντιμετωπίσει το σοβαρότατο πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα. Ο πρόεδρο και ο Πρωθυπουργός η κυβέρνηση στη Σρι το έχουν κάνει πρώτη κρατική προτεραιότητα. Πρέπει να τονίσω ότι η καλή συνεργασία μεταξύ κρατών, η μεγαστή συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος όχι μόνο στη Σρι αλλά και παντού στον κόσμο είναι ε, σοβαρότατη ανάγκη. Μόνο με τη διεθνή υποστήριξη μπορούμε να καταπολεμήσουμε τα καρτέλ των ναρκωτικών και άλλε εγκληματικέ δραστηριότητε. Η κυβέρνησή μου έχει καλέσει όλε τι χώρε συμπεριλαμβανομένων των εταίρων μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μας συνδράμουν προκειμένου να μπορέσουμε να εξαλείψουμε το φαινόμενο αυτό καθώς και τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και άλλες διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες ώστε να αποκατασταθεί η κοινωνία απαλλαγμένη από ναρκωτικά και η δημόσια τάξη που να προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μπορείτε να συνεισφέρετε κι άλλο στην οικονομική υποστηρίξη της χώρας μας. Γι' αυτό καλούμε τη διεθνή κοινότητα με τεχνική τεχνο, ε, ε, υποστήριξη και ό,τι τεχνογνωσία μπορεί να συνδράμε τη Σρι για να επιβάλλει σωστά τον νόμο και να υποστηρίξει και τις δικαστικές αρχές για να αντιμετωπίσουμε το κρίσιμο αυτό ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Ελπίζουμε να λάβετε ήδη κάποιες κατευθυντήριες γραμμές εδώ στο συνέδριο από πολιτικούς ηθήνοντες και υπουργούς. Θα ήθελα τώρα να στραφώ προς τον κύριο Γκακοσό που είναι υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Κογκό που κατέργησε στο σύνταγμα του 2015 τη θανατική πίνη. και μάλιστα γνωρίζουμε ότι η χώρα σας ε, κάνει κάποια διαβήματα προκειμένου να κυρώσει και το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο του Διεθνού Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Έχετε κάποια ανακοίνωση που να μας κάνετε σήμερα σχετικά. Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, κυρίες και κύριοι πρεσβευτέ, όντως η Δημοκρατία του Κονγκό το Σύνταγμα που υιοθετήθηκε με δημοψήφισμα τον Οκτώβριο του 2015 κατήργησε τη θανατική ποινή. Οπότε αυτή τη στιγμή η χώρα μου καλείται να κάνει ένα ακόμη βήμα σε αυτή τη μακρά πορεία προκειμένου να δώσει πλήρως νόημα στο δικαίωμα στη ζωή. Ένα δικαίωμα που είναι αμετάκλητο, όπως αναφέρθηκε και καταχειρώνεται και περιχαρακώνεται στο άρθρο 3 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο σημερινό 7ο συνέδριο ήρθα να επαναλάβω τη δέσμευση της χώρας μου να καταστήσει μία αντιστρέψιμη την κατάργηση της θανατικής ποινής ε, σφραγίζοντας την σε ένα δικαιικό σύστημα που τη θέτει στο απειρόβλητο των κυβερνητικών αλλαγών και των πολιτικών συγκυριών ή οποιονδήποτε σκαμπανεβασμάτων. Σε περιφερειακό επίπεδο την ίδια πυγμή και αποφασιστικότητα έχει και το Κονγκό που είναι υπέρ της έγκρισης από την Αφρικανική Ένωση του σχεδίου συμπληρωματικού πρωτοκόλου στον Αφρικανικό Χάρτη Δικαιωμάτων των Ανθρώπων και των Λαών που αφορά την κατάργηση της θανατική ποινή και σε διεθνέ επίπεδο, στο διεθνέ προσκήνιο. Από το Δεκέμβρη του 2007 η χώρα μου συστηματικά υπερψηφίζει όλα τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με στόχο να θεσπιστεί ένα παγκόσμιο δικαιοστάσιο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της θανατικής ποινής και υπερψηφίσαμε και το ψήφισμα για το μορατόριο όλα τα ψηφίσματα για το μορατόριο μεταξύ 2008 και 2014. Η κύρωση του δεύτερου προαιρετικού πρωτοκόλου στο Διεθνέ Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα θα είναι για τη χώρα μου το επιστέγασμα μιας ε, μακράς μάχης και πορείας που στόχο έχει να προτάξει για πάντα εναντί οποιοδήποτε άλλων αγαθών το δικαίωμα στη ζωή. Και μάλιστα ε, έχουμε καταργήσει το γνωστό νόμο της αντεκδίκησης των οφθαλμών αντιοφθαλμού που ουσιαστικά μας παραπέμπει σε κάποια ζωώδη αίσθηκτα και πολύ αρνητικές πτυχές της ανθρώπινης φύσης. Τον Οκτώβριο του 1982 είχαμε τις τελευταίες εκτελέσεις σε θανατική ποινή στο Κονγκό για δύο ανθρώπους που είχαν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Έκτοτε ακολουθήσαμε μία βολονταριστική πολιτική υπέρ της κατάργησης ε, και μάλιστα τη συνέχισε με πυγμή ο εξοχότατος πρόεδρος ε, της Δημοκρατίας του Κογκό, ο κύριος Ντένις Σασόν Γκεσό. Όπως σας είπα, 33 χρόνια έχουν περάσει από το 1982 και σε όλη αυτή την περίοδο δεν εφαρμόσαμε ουδέποτε την εσχάτη των ποινών. Και μάλιστα αυτό το μακροχρόνιο δικαιοστάσιο τελικά έπεισε την πλειοψηφία των συμπολιτών μου για την αναποτελεσματικότητα της θανατικής ποινής και την επιτακτική ανάγκη να την καταργήσουμε. Κάτι που τελικά καθαγιάστηκε, κατοχυρώθηκε, καταξιώθηκε στο Σύνταγμά μας της 15ης Οκτωβρίου του 2015, όπως σας είπα προηγουμένως. Μάλιστα το Σύνταγμα αυτό θεωρείται ιδιαίτερα πρωτοπόρο. Πρόκειται για ένα Σύνταγμα που είναι ένα σύνταγμα που καταργεί τη θανατική ποινή και ανοίγει μια νέα εποχή για τη χώρα μου. Και τέλος, κάποιος προλαλή σας μίλησε για το φίλο Ρομπέρ Μπαντεντέρ. Θυμάμαι ότι το Σεπτέμβριο του 1981 εκφώνησε την ομιλία του στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και είπε μεταξύ άλλων ότι όσοι πιστεύουν στην αποτρεπτική αξία της θανατικής ποινής αγνοούν την ανθρώπινη αλήθεια. Το πάθος του εγκληματία δεν θα το σταματήσει ο φόβος του θανάτου, όπως και άλλα πάθη δεν παρεμποδίζονται από κάτι τέτοιο και εκείνα τα πάθη είναι και πολύ πιο ευγενή. Αυτά είπε ο Ρόμπερ Πατεντέρ. Πώς λοιπόν να μην διαλογιστούμε σε αυτά τα βαρισίμαντα λόγια του Ρομπέρ Μπατεντέρ. Τόσο σοφά λόγια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη δέσμευσή σας κατά του νόμου του οφθαλμών οφθαλμού Ευχαριστώ που αναφέρετε τον κύριο Μπαντέντερ. Δεν είναι εδώ ε, μαζί μας, αλλά στο τέλος των εργασιών μας θα ακούσουμε ένα μήνυμα. Δεν είναι εδώ για λόγους υγείας. Καλημέρα σε ε, εξακό. Είστε Υπουργό Δικαιοσύνη τη Γουινέα, η οποία κατρίσει το 2016 θανατική ποινικά την ψήφο στη Γενική Σέλευση των Ηνωμένων Εθνών για ένα παγκόσμιο δικαιοστάσιο. Οι εκπρόσωποι σα απέσχουν. Του κράτου σα ε, σκοπεύει να επικυρώσει αυτό το δεύτερο πρωτόκολλο που έχει να κάνει με τα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. αξιολογικοί συνομιλητές. Καταρχάς, σα ευχαριστώ για τη δυνατότητα που δίνεται στην Δημοκρατία της Γουινέα να τονίσει τη δέσμευσή τη και την πρόοδο, πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ε, μάχη κατά της θανατική ποινής. Η Γουινέα ενέκρινε μία ιδιαίτερη μέθοδο. Η θανατική ποινή δεν έχει επισήμως καταργηθεί, αλλά τον Απρίλιο του 2016 Καταργήσαμε την θανατική ποινή, δηλαδή δεν αναφέρεται στο νέο μας ποινικό κώδικα. Η πλειονότητα των κατοίκων μας και η πολιτική και ορισμένες κοινωνικές τάξεις ε, εκφράζονται υπέρ της θανατικής ποινής λέγοντας ότι όταν υπάρχουν ειδικά φαινόμενα βίας τότε δικαιολογείται, γιατί έχουμε τέτοια φαινόμενα στη χώρα. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν αυτή τη μέθοδο. Πρώτα απ' όλα καταργήθηκαν τα ειδικά δικαστήρια και δώσαμε ποινικέ αρμοδιότητες ε, στα πρωτοδικεία. Έτσι τα 30 τέτοια πρωτοδικεία ε, ασχολούνται και με ποινικέ υποθέσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν τέτοια προδικεία ε, εύκολα να επιβάλλουν θανατικές ποινές. Και ενώπιον των κοινοβουλευτικών δώσαμε παραδείγματα που δείχνουν πώς έχει η κατάσταση και παρά τις πολιτικές διαφορές του κοινοβούλιο μας ομόφωνα εγκρίθηκε ε, αυτή η προσπάθεια. Τονίσαμε ότι ένας καινοτόμος ποινικό κώδικας δεν μπορούσε να περιέχει τη θανατική ποινή. Και εισακούστηκε αυτό το επιχείρημα. Έτσι λοιπόν από μορατόριουμ στην πράξη, γιατί οι τελευταίες ε, εκτελέσεις έγιναν το 2002, με το 2002 μέχρι το 2018 ήμασταν σε αυτή την κατάσταση, ναι μεν υπήρχαν 10 θανατοποιητέ στι φυλακέ δεν είχαν εκτελεστεί, αλλά με τον Απρίλιο, με το νέο ποινικό κώδικα τον Απρίλιο του 2016, δεν αναφέρεται πλέον η θανατική ποινή και οι ποινέ του μετετράπησαν σε ισόβια κάθριξη. Γιατί υιοθετήσαμε αυτή την ε, προσέγγιση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την ειδική κατάσταση σε κάθε χώρα. Βεβαίω, η αρχή της κατάργησης θανατικής ποινής ε, είναι βασική. Είναι μια πορεία ανεπίστρεπτη. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Αλλά ως πολιτικοί έχουμε κάποια ευθύνη. Η ευθύνη είναι να πείσουμε και την κοινή γνώμη και την ε, τάξη που λαμβάνει τις αποφάσεις για να μην υπάρξουν αντιφάσεις. Αυτό επιλέξαμε λοιπόν στην πράξη Μορατόριουμ για 15 χρόνια, τώρα μορατόριουμ και νομικό. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά μεταξύ της κατάργησης και το de jure moratorium που έχουμε στη Γουινέα. Αργότερα ένα απλό νομοθέτημα θα επιτρέψει στους βουλευτές μας να επικυρώσουν και επισήμως αυτή την κατάργηση. Η εικόνα που πολύ συχνά δίνω, καταλήγοντας, το είπα και στο Αμπιτζάνο που ήσασταν παρόντες ορισμένοι. Έχουμε ένα τριόροφο κτίριο που θέλουμε να φτιάξουμε. Το ισόγειο είναι οι χώρες που εφαρμόζουν ε, τακτικά την ποινή του θανάτου. Είναι μεγάλες ε, δημοκρατικές χώρες, ε, δεν θα τις αναφέρω, αλλά τις γνωρίζετε. Στον πρώτο όροφο έχετε τις χώρες που έχουν στην πράξη εφαρμόσει μορατόριο όπως η χώρα μου μέχρι το 2016 ναι μεν ε, οι δικαστές μπορούσαν να ε, καταδικάσουν εις θάνατον και ναι μεν δεν εκτελούντο αλλά έμεναν ως θανατοποιητές ειδικές πτέρυγες και μπορεί κάποια αλλαγή στην πολιτική κατάσταση να οδηγήσει στην εκτέλεσή τους. Λοιπόν, η, το de facto moratorium μπορεί να είναι επικίνδυνο. Ο δεύτερος όροφος είναι το de jure moratorium που αφαιρεί τη δυνατότητα αυτή από τον ποινικό κώδικα, άρα κανείς δικαστής δεν μπορεί να καταδικάσει θάνατον. Και για τους θανατοποινήτες υπάρχει μετατροπή των ποινών σε ισόβια. Στην περίπτωση της Γουινέας ε, η ελάχιστη ποινή που πρέπει να ε, τους επιβληθεί είναι 30 χρόνια, δηλαδή η ελάχιστη ε, διάρκεια της φυλάκισης. Και Κάποιες πιο ε, θαραλές χώρες όπως τη Μπουργκίνα Φάσο οι φίλοι μου με νόμο κατήργησαν επισήμως. Η διαφορά ανάμεσα σε εμά και σε όσους επισήμως κατήργησαν, κατά τη γνώμη μου, είναι μικρή. Απλώς λαμβάνουμε υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε χώρας. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή η πορεία είναι ανεπιστρεπτή. Ήθελα λοιπόν να σας περιγράψω την ε, πορεία της ε, χώρας μου, της Γουινέας. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει ηρεμήσει. Και βεβαίως χρειάστηκε να πείσουμε κάποιους ε, βουλευτές. Και τους είπαμε ότι πρέπει να το καταλάβουν, δεν μπορεί να υπάρχει και στα κείμενα. Και έχει γίνει αποδεκτή αυτή η κατάσταση πλέον. και γι' αυτό πολύ σύντομα θα υποβάλουμε ένα νομοσχέδιο. Άρα απαντώ στην ερώτησή σας επισήμως λέω ότι ναι είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε αυτό το δεύτερο πρωτόκολλο για την επίπτωση στα πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα και να το υποβάλουμε αυτό το πρωτόκολλο στην Εθνοσυνέλευση για επικύρωση. Ευχαριστούμε για αυτά τα καλά νέα, ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις σε σχέση με την ε, αναθεώρηση του ποινικού σα κώδικα. Το είπατε, κάθε, χρόνο, κάθε χώρα χρειάζεται τον χρόνο τη, κάθε χώρα έχει τι ιδιαιτερότητέ τη. Ε, σα αφήνουμε λοιπόν το χρόνο για να συνηθίσετε και τη γενική γνώμη τη χώρα σα στην αλλαγή. Τώρα, θα στραφώ στον Υπουργό ε, τη Μπουρκίνα Φάσο. Ε, είπατε κι εσεί ότι πρωτοπόρησε η ε, Μπουρκίνα Φάσο καταργώντα από το δικαστικό τη σύστημα τη θανατική ποινή. Και έγινε η πρώτη χώρα τη περιοχή που το έκανε αυτό. Συγχαρητήρια λοιπόν κύριε Μπάκορο. Ε, ωστόσο, η αφοσίωσή σα στον αγώνα μα δεν ε, σταματάει εκεί. Μπορείτε να μα πείτε περισσότερα. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι Υπουργοί, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών, θα μου επιτρέψετε εξ ονόματο τη αντιπροσωπεία μου να εκφράσω τι θερμέ μου ευχαριστίε προ το Βέλγιο, το Ευρωκοινοβούλιο και την ε, μη κυβερνητική οργάνωση όλοι μαζί κατά τη θανατική ποινή που προσκάλεσαν την Πορκίνα Φάσο σε αυτή την σημαντική εκδήλωση. Η χώρα μου ε, εκφράζει την ευχαρίστηση που συμμετέχει σε αυτό το παγκόσμιο συνέδριο και μαζί με όλου του συμμετέχοντε μπορεί να μοιραστεί την εμπειρία τη για το θέμα τη κατάργηση τη θανατική ποινή. Θεωρώ σημαντικό να ε, θυμίσω ότι ο δυναμικό χαρακτήρα του κινήματο για την κατάργηση τη θανατική ποινή στην Πορκίνα Φάσο απλώ διατηρήθηκε ακόμη και αν ο δρόμο ήταν και ε, δυσχερή λόγω ε, της αντίστασης της κοινής γνώμης ε, στο θέμα αυτό, παρά τον ενθουσιασμό ορισμένων την δάδα της πρόοδου την κράτησαν πολλοί πολιτικοί εκπρόσωποι, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και άλλοι συμμετέχοντες σε μη οργανώσεις ε, της χώρας και από τη διεθνή κοινότητα, ιδίως του ICP. Έτσι καταφέραμε να προχωρήσουμε και να αλλάξουμε τα πράγματα από την οθέτηση του συντάγματος το 1991. Έκτοτε η χώρα προχώρησε στη δημιουργία ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου που βασίζεται στην δημοκρατική άσκηση των ε, ατομικών και συλλογικών ομαδικών δικαιωμάτων. Έτσι ε, κυρώσαμε τα διάφορα περιφερειακά και διεθνή εργαλεία ιδιαίτερη σημασία, ε, όπω το μορατόριο για τη θανατική ποινή, που μα επέτρεπαν να δημιουργήσουμε ακριβώ αυτό το ελεύθερο δημοκρατικό καθεστώ. Έτσι, ε, βλέπαμε ότι η διατήρηση τη θανατική ποινή στην ε, εθνική νομοθεσία θα δημιουργούσε προβλήματα στη συμβατότητά του με τι διεθνεί μα δεσμεύσει και το σύνταγμα τη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική τάξη τη Μπουρκινας Φάσο διοργάνωσε προσπάθειες, συζητήσεις, διαβουλεύσεις ε, και εκστατείες ευαισθητοποίησης προς όλες τις κοινωνικο-οικονομικές ε, ομάδες της χώρας για να τους ε, ευαισθητοποιήσουμε και να τους ενημερώσουμε. Με δύο νόμους προχωρήσαμε τα τελευταία χρόνια στην κατάργηση της θανατικής ποινής και των μεσανιστήριων που τελικά οδήγησαν στην πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής ιδίως το 2015 με τις 7 περιφερειακές εκστρατείες σε περιφερειακό επίπεδο για την ε, ε, κατάληξη της θανατικής ποινής και για την ενημέρωση των δικαστικών λειτουργών, την προάσπιση των ε, τοπικών φορέων, την προάσπιση της ανεξιθρησκείας όσων είναι ηγέτες της κοινή γνώμης, και ούτω καθεξής. Με το σχέδιο του νόμου, του νέου συντάγματος μάλλον στο εδάφιο 5, προβλέπεται ότι δεν μπορεί να ασκηθεί ποτέ και να εφαρμοστεί η θανατική ποινή. Θα εγκριθεί το Μάρτιο το νέο σύνταγμα. Ωστόσο, παρά τις κοινωνικές αυτές ε, καταστάσεις, ορισμένα κοινωνικά γεγονότα και κατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή νοτίως της Σαχάρας έχουν ε, φέρει σε δύσκολη ε, θέση την, ε, το ολοκίνημα της κατάργησης. Οι προσπάθειες ευαισθητοποίησης, πέρμαχοι της κατάργησης και όσοι έχουν δεσμευτεί στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής δεν κατάφεραν τελικά να καταλήξουν σε μια πλήρη συμφωνία. Επειδή λοιπόν δεν υπήρχε συνένεση σε σχέση με το θέμα τη κατάρριξη τη θανατική ποινή, η κυβέρνησή μα αποφάσισε να καταγράψει τη χώρα μα στο συνολικό πίνακα και στο να ε, ε, τοποθετήσει στο τοπίο των χωρών που έχουν προχωρήσει στην πλήρη κατάργηση. Γι' αυτό λοιπόν η κατάργηση της θανατικής ποινής προβλέφθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών στην συνεδρίασή του 14 Μαρτίου 2018 με το νομοσχέδιο για την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 31 Μαΐου 2018. Έτσι ε, μπορέσαμε να καθιερώσουμε την κατάρριξη της θανατικής ε, ποινή στην πουρκινα Φάσο. Όπως βλέπετε αυτό το πετύχαμε από τις 31 Μαΐου 2018 χάρη στην στενή συνεργασία των κρατικών αρχών της χώρας ε, και την υποστήριξη που είχαμε από τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών. Ε, Βεβαίω, το τελικό ε, καθοριστικό ε, στοιχείο και όπλο για όλο αυτόν τον αγώνα ήταν η πολιτική βούληση στη χώρα μου. Και θα ήθελα με αυτό να κλείσω, προσκαλώντα τι χώρε που ακόμα αντιστέκονται στην κατάρριξη τη θανατική ποινή να εκφράσουν χειρά την βούλησή του να προχωρήσουν σε αυτόν τον δρόμο και θα σα καλωσορίσουμε και εμεί στην ομάδα των χωρών που συμμετέχουν στην κατάρριξη τη θανατική ποινή παγκοσμίω. Σας ευχαριστούμε κύριε Βαυρό και ευχαριστούμε για την έκκληση σας προς χώρες που εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη θανατική ποινή και ευχαριστούμε και τη δέσμευσή σας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αναγγείλατε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Αμπουμπακάρ Ταμπαντού, Γενικός Εισαγγελέας και Υπουργός Δικαιοσύνης της Γκάμπια. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Το 2018 η Γκάμπια κύρωσε το δεύτερο προαιρετικό πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινή. Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την κατάργηση της θανατικής ποινή στην Γκάμπια. Σας ερωτούμε λοιπόν πότε ε, θα υιοθετήσετε και την κατάλληλη νομοθεσία για να τηρήσετε τις διεθνείς σας δεσμεύσεις ως προς το θέμα της κατάργησης θανατικής ποινή. Σας ευχαριστώ, εξοχότητες ε, ε, διακεκριμένη καλεσμένη, Θα ήθελα να σταθώ στο πρωτόκολλο. Η θανατική ποινή καταργήθηκε το 1993 στην Κάμπια, αλλά επανήλθε το 1995 μετά από ένα στρατιωτικό πραξικόπημα που έλαβε χώρα το 1994. Οι λόγοι που δόθηκαν από την στρατιωτική χούντα για την επαναφορά της θανατικής ποινής τότε ήταν, και παραθέτω εδώ, μια από την κατάργηση της θανατικής ποινής στην Κάμπια ε, παρατηρήσαμε μια σταθερή αύξηση των ανθρωποκτονιών και των περιπτώσεων προδοσίας. Αν δεν ελεγχθεί αυτή η κατάσταση μπορεί να εκφυλιστεί και να οδηγήσει σε μια κατάρρευση του νόμου και της τάξης. Αυτά ισχυρίστηκε τότε η στρατιωτική χούντα για την επαναφορά. Δεν υπήρχαν όμως ε, πραγματικές αποδείξεις και τεκμήρια που να στοιχειοθετούν αυτό το επιχείρημα. Ήταν ένα απλό πρόσχημα. Και μάλιστα ε, η αύξηση των ανθρωποκτονιών ήταν απόρρια των δράσεων της στρατιωτικής χούντας. Ε, ένα νέο σύνταγμα εγκρίθηκε το 1997 στην Κάμπια που εγγυάται το δικαίωμα στη ζωή. Το ίδιο Σύνταγμα διατηρεί τη χρήση της θανατικής ποινή για διακεκριμένα εγκλήματα, αλλά προβλέπει ότι, μέσα σε 10, ότι μετά από 10 χρόνια ή μέσα σε 10 χρόνια από τη θέση σε ισχύ του νέου συντάγματος, η Εθνική Συνέλευση της Γκάμπια θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα ή θα προβεί σε ολοσχερή κατάργηση της θανατικής ποινής στη χώρα. Κάτι που δεν έγινε ποτέ. Οπότε η θανατική ποινή εξακολουθεί να είναι ε, επιλογή, πιθανότητα, αλλά δεν έγιναν ε, καθόλου εκτελέσεις μέχρι τον Αύγουστο του 2013, οπότε εννέα άτομα κρατούμενοι στη φυλακή Μάιλ 2 εκτελέστηκαν και μάλιστα πολλοί ισχυρίστηκαν ότι ε, εκτελέστηκαν με κατάφορη παραβίαση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Μετά την αλλαγή στην κυβέρνηση στην Κάμπια το Δεκέμβριο του 2016, ένα δικαιοστάσιο στην εφαρμογή της θανατικής ποινής επευλήθη από το Φεβρουάριο του 2018 και όλες οι θανατικές καταδίκες έχουν έκτοτε μετατραπεί σε ισόβια τον Αύγουστο του 2018. Ακολούθησε, ε, κάτι που ακολούθησε ε, το Σεπτέμβριο του 2017 την κύρωση από την Γκάμπια του δε, της Γκάμπιας του δεύτερου Πρακτικού πρωτοκόλου του Διεθνού Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σε ό,τι αφορά την κατάργηση θανατικής ποινή. Παρ' όλα αυτά, το θέμα της θανατικής ποινή είναι συνταγματικό ζήτημα για την Γκάμπια. Οπότε η κατάργηση της θανατικής ποινή προϋποθέτει μια συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια ε, αξιολόγηση του συντάγματος και μια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης και όπως αναμενόταν έγιναν εκτεταμένες συζητήσει επ' ευκαιρία αυτής της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η νέα κυβέρνηση της Γκάμπια απερίφραστα στηρίζει την ολοσχερή κατάργηση της θανατική ποινή στην πατρίδα μου. Ευχαριστώ. Thanks, Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Οι κυβερνήσει μπορούν να ηγηθούν τη κοινή γνώμη για την κατάργηση Στηρίζουμε ε, την τόλμη τη κυβέρνηση προσπαθεί να αναθεωρήσει το Σύνταγμα και ελπίζουμε σύντομα να καταργηθεί η θανατική ποινή. Σήμερα έχουμε επίση και τον Υπουργό Δικαιοσύνη του Μαρόκου, Μαμέντου Ζάρ. Καλημέρα σα. Σα παρακαλώ να μα πείτε πώ αναγράφει το δικαίωμα στη ζωή στο νέο Σύνταγμα, καθώ και τι πολλέ ε, δηλώσει του βασιλέως ε, Μοχάμεντ Έκτου υπέρ τη κατάργηση. Ποια θα είναι τα πρώτα βήματα και πότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα καταργηθεί η θανατική ποινή. Ευχαριστώ κυρία πρώτα Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Έχω πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη συγκίνηση που συμμετέχω σε αυτήν τη διακεκριμένη εκδήλωση. Και υπενθυμίζω ότι το βασίλειο του Μαρόκου υπό την ηγεσία του βασιλέως ε, Μοχάμεντ Έκτου θέλει να δημιουργηθεί ένα κράτος δικαίου, μια δημοκρατική πολιτεία με πλήρη σεβασμό όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως ε, τονίσατε, χάρη σε ένα εθνικό διάλογο καταφέραμε κατά την σύνταξη του νέου συντάγματος να βάλουμε το άρθρο 20 που αναφέρεται το δικαίωμα στη ζωή που είναι το πρώτο αρχικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Ο νόμος προστατεύει αυτό το δικαίωμα αυτή η σαφής αναφορά είναι πολύ σημαντική. Είναι μια σημαντική εγγύηση του πόσο θέλουμε να προχωρήσουμε. Η χώρα μου έχει υιοθετήσει μια στρατηγική μη εφαρμογή των θανατικών ποινών. Σας διαβεβαιώ ότι καμία εκτέλεση δεν έχει γίνει από το 1993 και εντεύθεν. Και καμία εκτέλεση δεν θα επιτραπεί αυτή η στρατηγική <clears throat> μη εφαρμογή της θανατική ποινή είναι ακριβώ αποτέλεσμα του εθνικού διαλόγου γύρω από το θέμα αυτού. Και για λόγους διεθνούς και περιφερειακής ε, συγκυρίας οι κοινωνίες μας ε, διατρέχονται από ένα κύμα συντηρητισμού που παίζει μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση της στρατηγικής μας για τη δημοκρατία. Το θέμα αυτό δημιουργεί συγκρούσεις. Γίνεται λοιπόν μία συζήτηση. Η στρατηγική μας προσπαθεί να περιορίσει νομοθετικά. Έναντι του Κοινοβουλίου θα παρουσιάσουμε ένα νέο σχέδιο ποινικού κώδικα που θα περιορίσει τον αριθμό των περιπτώσεων και υποθέσεων ε, για τις οποίες μπορεί να επιβληθεί η θανατική ποινή. Από 31 αδικήματα που μπορούν να επιφέρουν τη θανατική ποινή, έχουμε μειώσει ιδιαίτερα την περίπτωση μόνο σε περιπτώσεις ε, γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εσχάτης προδοσίας. Όπως είπα και χθε στην κυρία Πιλάη, είμαι αισιόδοξο. Ελπίζω ότι η συζήτηση αυτή θα οδηγήσει στην πλήρη κατάργηση στο Μαρόκο. Είμαστε σε σταδιακή θετική πορεία. Πραγματιστική βέβαια. Εδώ και πάνω από 40 χρόνια και με το διάλογο που θα ξεκινήσει σύντομα στο Μαρόκο και με το δυναμισμό της κοινωνίας των πολιτών ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια συνένεση γύρω από την προσπάθεια αυτή. Έχω κάθε εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της χώρας μου να αναγγείλει καλά νέα σύντομα για το θέμα αυτό. Καταλήγω με αυτό το αισιόδοξο πνεύμα αποτείοντας θερμό φόρο τιμής στην κοινωνία των πολιτών, στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι και εδώ παρόντες, που αντιμετωπίζουν αυτό το κύμα συντηρητισμού αποφασιστικά, όρθιοι στηρίζουν αυτήν την ευγενή προσπάθεια και τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ουζάρ, ευχαριστώ που υπενθυμίσατε για μια φορά το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή τη μάχη. Ξέρουμε ότι αυτή η μάχη και ο διάλογος είναι ιδιαίτερα έντονος και θέλουμε να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια στην πράξη κατάργησης της θανατικής ποινής. Ευχαριστώ τους Υπουργούς που μας δώσατε ένα απολογισμό της κατάστασης της χώρας σας και τόσα καλά νέα. Αλλά τι σημαίνει να είναι κανείς θανατοπινίτες. Οι φυλακισμένοι πώς ζουν και πώς ε, διατηρούν την ανθρώπινη επαφή με τους άλλους ε, φυλακισμένους. Ο Ντουμέι Τουσάνι πέρασε 20 χρόνια στο Τένεση, στο, στην πτέρυγα των θανατοποιητών για ένα έγκλημα που δεν είχε διαπράξει στη φυλακή ξεκίνησε να μαθαίνει να ζωγραφίζει και έτσι μπόρεσε να εκφράσει στην ε, απομόνωση την, ε, ε, να, να εκφράσει την άποψή του και σήμερα θα μας παρουσιάσει ένα έργο του. Τον ευχαριστούμε. Uh, uh, Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που το παρουσιάσατε αυτό εδώ στο κέντρο του Εμικυκλίου. Σας ευχαριστώ που το δεχτήκατε καταρχάς. Και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Μου φαίνεται απίστευτο που βρίσκομαι εδώ. Όπως ακούσατε, Συνολικά πέρασε 20 χρόνια στη φυλακή. Στο θάλαμα με θανάτων του Τενεσί. Για ένα δίκημα που είχε δικαστή από νωρί, αλλά το τεκμήριο αθωότητα στην περίπτωσή μου καταρρίφθηκε πλήρω, γιατί οι κατηγορίε εναντίον μου ήταν χαλκευμένε όλε και τέλο πάντων δεν κατάφερα ποτέ να αποδείξω την αθωότητά μου. Το κράτο με καταδίκασε. Εάν δείτε τι είναι η πηγή του πολιτισμού, Πρέπει να πάτε πολύ μακριά, στην προϊστορία, πριν χιλιάδες χρόνια από κόσμο ζούσαν στις σπηλιές. και έβαζαν το χέρι του στο τείχομα της σπηλιάς και με χρώμα γύρω έφτιαχναν ένα σχήμα. Εγώ λοιπόν, όταν βρέθηκα να κάθομαι σε τέτοιο κελί ε, για μελοθανάτους και να βρίσκομαι σε μια παρόμοια κατάσταση, θυμήθηκα τι είχα μάθει ως σχολείο. Δεν είχα κανένα ιδιαίτερο σχολικό ενδιαφέρον. Αλλά το μόνο που μου άρεσε να κάνω στη ζωή μου, πραγματικά, και αυτό μου την έσωσε τη ζωή μου, ήταν το λάδι. Ε, έτσι κατάφερα να σώσω τη ζωή μου και υπό κάθε περίσταση σε κάθε διαφορετικό ε, περιστατικό που ζούσα, ήταν δύσκολο να διατηρήσω τη διάθεσή μου για επιβίωση. Αλλά αυτό εδώ που έφτιαξα για αυτή την εκδήλωση, βλέπετε τι απεικονίζει. Έναν ε, άνθρωπο να κάθεται στην ηλεκτρική καρέκλα. Και γι' αυτό έχω βάλει και αυτά τα καλώδια στο κεφάλι του, γιατί έτσι γίνεται η εκτέλεση. Τέλος πάντων αυτό είναι κάτι που βρίσκεται, γίνεται ακόμα μόνο στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάποιες άλλες χώρες στον κόσμο. Και ήμουν τυχερός που πήγα και στο έκτο συνέδριο, στο Όσλο, ε, και στο τέλος της εκτέλεσης είχαμε βρεθεί τρεις Βάλαμε τα χέρια μας και το αποτύπωμά μας σε διάφορα σημεία. Ήταν πολύ ισχυρό αυτό που κάναμε τότε. Γιατί για μένα, εμείς που είμαστε κατά αυτές της αδικίας, πρέπει πάντα να αφήνουμε το αποτύπωμά μας παντού. Αν δεν υπήρχαν άνθρωποι σαν και εσά που μα βοηθάνε και είναι κατά τη θανατική ποινή, δεν θα ήμουν εδώ σήμερα. Α, εσείς μου δώσατε ελπίδα. Εσείς μου επιτρέψατε να σηκώνομαι κάθε πρωί και να έχω ελπίδα. Να κάνω ό,τι μπορώ για να προχωρώ. Ακόμη και αν ήμουν απεγνωσμένος. Σηκωνόμουν όπως σας είπα. Σας είπα το, το λάδι, τα, η ζωγραφική με το λάδι για μένα, όπως σας είπα δεν με ενδιέφερε παλιότερα. Πώ τα κάλυψα, πώ μπορώ να ζωγραφίσω. Ήταν κάποιο άλλο θανατοποιητή που κατόπιν εκτελέστηκε. Αυτό τι ήταν καλλιτέχνη. Και του είπα, κάνε μου μια ζωγραφιά να στείλω στη μητέρα μου. Όταν την τελείωσε, βέβαια δεν μου μοιάζε καθόλου. Δεν έμοιαζε με τίποτα. Κάθομαι εκεί πέρα, σε αυτό το περιορισμένο χώρο του κελιού μου και είπαμε, εγώ θα μπορούσα να το έχω κάνει καλύτερο και να μην τον πληρώσω. Και ευτυχώς... Η μητέρα μου δεν την είδε ποτέ αυτή τη ζωγραφιά που έκανε ο άλλο. Ήταν δύο χρόνια που ήμουν φυλακή. Γιατί η μητέρα μου δυστυχώ σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό ατύχημα. Κοιτάξτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, είναι δύσκολο να τα σκεφτώ τα πράγματα. Μου έρχονται δάκρυα. Με συγχωρείτε, μου έρχονται δάκρυα όταν σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν ε, φυλακισμένο, σε οποιονδήποτε μπορεί να συμβεί, αλλά ιδιαίτερα στη φυλακή δεν ελέγχει τίποτα. Και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι, κοιτάξτε, έρχεται, έρχεται κάποιο στο κελί σου και σου λέει μπορεί να τηλεφωνήσει σπίτι σου. Όταν στο πούν αυτό, ξέρει ότι κάτι έπαθε κάποιο δικό σου. Κάτι σοβαρό πρέπει να συμβεί. Κάποιο πρέπει να πεθάνει για να σου δώσουν ένα δωρεάν τηλεφώνημα. Και όταν ήρθα στο κελί μου και μου είπανε έλα να πάρεις ένα τηλέφωνο κατάλαβα συνέχεια όταν βγαίνω από το κελί μου και μου λένε ότι έλα εμπρό, τι θα μου πει η μητέρα μου στο τηλέφωνο τι συνέβη σε ποιον και όταν πήγα κάτω μίλησα με την αδελφή μου που μου είπε ότι είχε σκοτωθεί η μητέρα μου και όταν μου το έλεγε δεν μπορώ καν να το καταλάβω, να το δεχτώ. Δεν άκουγα, δεν ήθελα να ακούσω αυτό που μου έλεγε. Ε, μετά από μερικά δευτερόλεπτα βέβαια τα ακούς. Τις πρώτες τρεις μέρες που μου το είπαν έκλαιγα συνέχεια. Αλλιώς προσπαθούσα να ξεφύγω από την πραγματικότητα, κουλουριασμένος. Τρει μέρες μετά εκεί ήμουνα στο κρεβάτι, δεν ήθελα να σηκωθώ, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Είδα τη μητέρα μου, σαφώς στα μάτια μου και μου είπε σήκω. Σηκώθηκα πάνω και έτσι τελείωσαν οι εφιάλτε. Δέχτηκα την πραγματικότητα. Μετά από αυτό κάθομαι στο κελί μου, τέσσερα πόδια επί εννέα, και κοιτάω αυτή την εικόνα, τη ζωγραφιά που ήθελα να της έχω στείλει. Και τότε κατάλαβα. Αφού μου είπε η μητέρα μου να σηκωθώ, κάθε φορά που έβλεπα αυτή τη ζωγραφιά, αυτό το πορτρέτο, έλεγα Σκέφτηκα πάλι αυτό το οποίο είπα όταν το πρώτο είδα. Γιατί να τον πληρώσω, εγώ θα την είχα κάνει καλύτερα. Τότε ακριβώς, τότε ανακάλυψα τις ελαιογραφίες. Και Μέσω της ζωγραφικής βρήκα την ελευθερία. Εκεί που ήμουν μέσα στο κελί μου βρήκα την ελευθερία. Και έτσι μάλιστα και άλλοι με προσέγγισαν όταν ήταν τις ζωγραφιές μου. Πραγματικά η ζωγραφική μου έσωσε τη ζωή. Γιατί μόνο τότε με είδαν από πιο κοντά οι άλλοι και κατάλαβαν ότι ήμουν στη φυλακή για κάτι που δεν είχα κάνει. Και αυτό σας λέω. Αυτό επέτρεψε και στην οικογένειά μου και σε άλλους που πάντα με στήριζαν, αλλά και σε άλλους ευρύτερα να έρθουν, να ακούσουν και να καταλάβουν όχι μόνο τι συμβαίνει σε μένα, αλλά και σε άλλους. Γιατί υπήρχαν και άλλοι δύο που ξέρω με βάση αυτά που μου είπαν και πραγματικά τους πίστεψα, ξέρω ότι ήταν στην ίδια περίπτωση με τη δική μου. Δεν είχαν κάνει το έγκλημα για το οποίο είχα καταδικαστεί. Και ξέρω αυτά τα άτομα που τώρα δεν είναι πια θανατοποινήτες γιατί τους έκαναν οι εισαγγελίες και η αστυνομία και οι δικαστές τα ίδια που είχαν κάνει και σε μένα. Και το πιστεύω αυτό. Είχαν πάθει τα ίδια με μένα. Αν δεις ε, πώς με είχαν αντιμετωπίσει εμένα, το είχαν κάνει και στα άλλα δύο αυτά άτομα που και αυτοί ήταν ε, φυλακισμένοι θανατοποινήτες. Όπως σας είπα, κοιτάξτε, είναι καταπληκτική αυτή η ευκαιρία από όταν ε, αποφυλακίστηκα να ταξιδέψω στον κόσμο, να εργαστώ και στη χώρα μου και όχι μόνο στη χώρα μου με νέα παιδιά, να προσπαθήσω να τα πείσω. Είναι τρομερό αυτό που μου έκανε η ζωγραφική. Είναι τρομερό, τρομερά δυνατό όταν προσπαθείς να έρθεις σε επαφή να πλησιάσεις ανθρώπους για διάφορα θέματα. Δουλεύω με νέα παιδιά, με τη ζωγραφική. Προσπαθώ να τους ενημερώσω. Δεν ξέρω πόσα ξέρετε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι φυλακές είναι τρομερή βιομηχανία. Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω ότι και πριν μπω φυλακή ήμουν καλλιτέχνη, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω αυτά που έκανα ω θανατοπινίτης. Αυτό λέω και στους νέους. Πρέπει να καταλάβουν. Πρέπει να καταλάβουν πώς λειτουργεί το σύστημα γύρω τους. Γιατί όπω σας είπα, το να κλείνουν ανθρώπου στη φυλακή είναι βιομηχανία εκατοντάδων εκατομμυρίων ετησίω. Και κοιτάξτε, οι άνθρωποι που είναι φυλακοί είναι όπως ε, εγώ και εσείς εδώ μέσα. Δεν είναι διαφορετικοί. Είναι καταπληκτική η ευκαιρία που μου δόθηκε γιατί θα μπορούσε να ε, αποφυλακιστώ και απλώς να γυρίσω στο σπίτι μου να προσπαθήσω να ξεχάσω. Αλλά έδωσα υπόσχεση στους άλλους φυλακισμένους όταν έβγαινα ότι όταν βγω θα υψώσω τη φωνή μου, θα προσπαθήσω να βοηθήσω γιατί ήξερα ότι άλλοι είχαν μιλήσει πριν για μένα. Άνθρωποι όπως εσείς. Άνθρωποι εσείς, εσείς με βγάλατε από τη φυλακή. Άνθρωποι που χωρίς να με ξέρουν αγωνίζονταν για μένα όσο ήμουν φυλακή. Κοιτάξτε, ό,τι μας πληγώνει στη ζωή ότι σε ρίχνει κάτω μπορεί να ε, σε βοηθήσουν άλλοι να ξανασηκωθείς να καταλάβεις ότι έχεις ε, και εσύ ευθύνη όταν βλέπεις κάποιον που τον έχει χτυπήσει η ζωή να προσπαθήσετε να τους πείτε σήκω μην χάνεις την ελπίδα όλα είναι δυνατά είμαι εδώ τώρα και πρέπει να σας πω ότι μακάρι να ήξερα πώς θα μπορούσα το πνεύμα που υπάρχει εδώ μέσα να το κλείσουμε κάπου και να το δώσουμε στα άτομα που είναι ακόμη μέσα. Σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Πρέπει να το συνεχίσουμε. you, Ευχαριστούμε, Ντούμε, που, μας, ε, που μοιράστηκες μαζί μας την προσωπική σου ιστορία και τα αισθήματά σου. Ελπίζουμε με τη συνεργασία μας να αλλάξουμε το σύστημα. Ε, ο τύπος του Μαρόκου ε, μιλά για το πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει στην προσπάθεια κατάργησης του θανάτου και μάλιστα το 1993 που έγινε η τελευταία εκτέλεση στο Μαρόκο δήλωσε την αντίθεσή του στη θανατική ποινή. Νούζα Σκάλι, επανειλημμένος υπουργό στο Μαρόκο, είναι σήμερα μέλος της ε, Επιστημονικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συνεδρίου για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Κυρία Νούζα Σκάλι, παρακαλώ έχετε το λόγο. Τι δύσκολο που είναι να παίρνει κανείς το λόγο μετά τη συγκλονιστική μαρτυρία του Ντούμ. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε, ίσα ίσα μας εμψύχωσε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Αγαπητοί υπέρμαχοι της κατάργησης της θανατικής Ποινή από τις πέντε υπήρους, αξιότιμοι συνάδελφοι, ε, νιώθω μεγάλη τιμή και προνόμιο που βρίσκομαι εδώ ενώπιον των 1500 υπερμάχων της κατάργησης θανατικής ποινής, αυτό το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο που οργανώνεται στις Βρυξέλλες την πρωτεύουσα της Ευρώπης και σήμερα πρωτεύουσα του κόσμου για την κατάργηση θανατικής ποινής και μάλιστα σε αυτό το συμβολικό χώρο, στην αίθουσα της Ολομέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συνοδιοργανωτές, τους χορηγούς της οργάνωσης, την οργάνωση Together ε, Against the ε, Death Penalty, τον κύριο Χαζάν, και τους εταίρους, ε, τους συνδιοργανωτές αυτού του σημαντικού παγκόσμιου συνεδρίου και να ευχαριστήσω την οργάνωση μαζί κατά της θανατικής ποινή για τις ε, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν υπέρ της κατάργησης παντού στον κόσμο και κυρίως στην Αφρική και στο Μαρόκο για την υλοποίηση του κοινού μας στόχου που είναι η καθολική παγκόσμια κατάργηση αυτού του ε, αιώνιου στίγματο της θηριωδία, όπω έλεγε ο Βίκτορ Γκό, για αυτή τη απάνθρωπης εξευτελιστική ποινή που είναι η θανατική καταδίκη. Η πορεία μα ε, προ την κατάργηση είναι αναπόδραστη. Ακολουθεί την πορεία τη ιστορία, το ρου της ιστορίας, στηρίζεται στι ανθρωπιστικέ αξίες, ε, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στο δικαίωμα τη ζωή. Και όπω μα έδειξαν αυτέ οι γλαφυρέ και εύγλωτε ομιλίε που ακούσαμε, Σίγουρα, χάρη σε αυτό το 7ο συνέδριο, οι καρδιές μας πάλλονται στον ίδιο ρυθμό. Θέλουμε να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτήν την αναποτελεσματική και διακριτική πρακτική και να αναπτύξουμε στρατηγικές παγκοσμίω για να επιταχύνουμε το ρου της ιστορίας προς την κατάργηση, την παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής και στα Ω μέλο τη Επιστημονική Επιτροπή, ε, είχα την τιμή να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία που έγινε χωρί αποκλεισμού για να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα του συνεδρίου με βάση τις προτάσεις τη οργάνωση ICPM και της ε, παγκόσμια Συμμαχίας κατά της θανατική ποινή. Έχουμε μια πολυεθνική πολυμελή εταιρεία που διαπνέεται κυρίως από τις αρχές ε, κατά της θανατική ποινής. Και η κυρία Σέινα ηγήθηκε των διαδικασιών και την συγχαίρω και την ευχαριστώ θερμά και σας μεταφέρω και τον θερμό χαιρετισμό της Επιστημονικής Επιτροπής. Έχουμε, πολλές, ε, έχουμε αυτή τη συνεδρία σήμερα, αλλά και πολλές ε, συναντήσεις έγιναν μέχρι, μέσα από το Skype. Επιστέχασμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι η σημερινή ημέρα, το σημερινό συνέδριο. Θέλουμε να διευρύνουμε τους τομείς και τις κατηγορίες ε, των πολιτών που θα λάβουν μέρος αυτή τη μεγάλη μάχη για την κατάργηση μαζί με τον ιδιωτικό τομέα που πρώτη φορά συμμετέχει σε ένα παγκόσμιο συνέδριο για την κατάργηση θανατικής ποινής. Η διακριτική εφαρμογή της θανάτικης ποινής εις βάρος των γυναικών είναι ένα νέο θέμα που μας προβληματίζει. Πολύ συχνά η διάκριση αυτή οφείλεται στο φαλοκρατικό πατριαρχικό σύστημα που εφαρμόζεται εις βάρος των γυναικών και η θανατική ποινή προστίθεται στις άλλες μορφές βίας ε, εις βάρος των γυναικών και υποτίθεται ότι ε, τιμωρεί υποδειγματικά ε, παιδοκτονία, μοιχεία ή άλλα εγκλήματα στο πλαίσιο του γάμου. Επίσης, πολλές φορές οι γυναίκες ε, καταδικάζονται στο όνομα της θρησκείας. Θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη σε κλήσεις μας για την κατάργηση, προωθώντας ε, ειρηνιστικό ανθρωπιστικό περιεχόμενο που σέβεται την ανθρώπινη ζωή σε όλες τις θρησκείες. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν και το συνέδριο. Θα πρέπει επίση να ενδιαφερθούμε για τις οικογένειες των καταδίκων και κυρίως για τα παιδιά. Αυτό είναι ένας καινοτόμο τρόπος για να διευρύνουμε το πεδίο των ε, ατόμων που θίγονται από την, κατα... από την θανατική καταδίκη ενό οικείου. Και αυτοί οι συγγενείς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στη γενική συζήτηση. Και έχουμε μαρτυρίες από μέλη της οικογένεια... οικογένειας των ε, καταδίκων, από δικηγόρους και ούτω καθεξής. Για 30 χρόνια είμαι ακτιβίστρια για την κατάργηση και είμαι υπερήφανη που κατάγομαι από την Αφρικανική Ήπειρο, την οποία λατρεύω. Και μετά την επιστροφή του Μαρόκου τον Ιανουάριο του 2017 ε, και με την επιστροφή του Μαρόκου στην οργάνωση αυτή χαίρομαι ιδιαίτερος. Ε, πιστεύω ακράδαντα ότι η Αφρική θα είναι η επόμενη ήπειρος που θα προβεί σε καταργήσεις, γιατί ε, οι περισσότερες χώρες Αφρικής ε, από τις 41 είναι de jure ή de facto ε, χώρες που έχουν καταργήσει το, τη θανατική καταδίκη. Και στην πατρίδα μου ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει πολύ χρόνες ρίζες. Περιλαμβάνει το δικαίωμα στη ζωή, τα θεμελιώδη δικαιώματα και σίγουρα το δικαίωμα στη ζωή κατοχυρώνεται και στο άρθρο 20 του Μαροκινού Συντάγματος της 1 η Ιουλίου του 2011 και εμψυχωμένοι από όλη αυτή τη δημοκρατική διαδικασία, δημιουργήσαμε το 26 Φεβρουαρίου του 2013 ένα κοινοβουλευτικό δίκτυο κατά τη θανατική ποινή στο Μαρόκο. Με πρωτοβουλία βουλευτών και διαπνεόμενη από οικουμενικές ανθρωπιστικέ αξίες ε, κατά της θανατική ποινή. Έχουμε ταυτόχρονα επίγνωση ε, του ρόλου των βουλευτών που είναι νομοθέτες και επίσης συμβολίζουν την κυριαρχία του έθνους. Η πρωτοβουλία μας στέφθηκε με επιτυχία χάρη στην υποστήριξη και της Μαροκινής Συμμαχίας κατά της θανατικής ποινής. Χαιρετίζω και τον πρόεδρο της οργάνωσης και με την βοήθεια της οργάνωσης μαζί κατά της θανατικής ποινής. Ε, έτσι, χάρη στην υπερκομματική προσέγγιση, είχαμε την υποστήριξη 240 βουλευτών από κόμματα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Και μάλιστα οργανώσαμε πολλά σεμινάρια και συμμετείχαμε και σε διεθνή συνέδρια κατά της θανατικής ποινής στη Μαδρίτη το 2013, στο Όσλο το 2015 και πρόσφατα το 2018 στο τρίτο περιφερειακό συνέδριο στην Αμπιτζάν κατά της θανατικής ποινής. Η εμπειρία μας ήταν άνευ προηγουμένου, πρωτοπόρα, καινοτόμα και υπόδειγμα παράδειγμα προ μίμηση για τι χώρε που δεν έχουν ακόμη καταργήσει τη θανατική ποινή. Πολλέ φορέ ε, νιώσαμε ότι ήμασταν κοντά στην επίτευξη του στόχου μα όταν το Εθνικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έθεσε την έκθεσή τη στο Κοινοβούλιο και έβαλε την κατάργηση θανατική ποινή ω ύψιστη προτεραιότητα των συστάσεων. Και χαιρετίζω την Αμήνα Μποαγέ, τη νέα πρόεδρο αυτού του Εθνικού Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μαρόκου, που μάλιστα παρούσα στην Ομίγυρη, αλλά και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Φόρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έγινε στο Μαρακέ ε, τον Νοέμβριο του 2014, ε, διατρανώσαμε τη δέσμευσή μα και εκεί χιλιάδε ακτιβιστέ και ακτιβίστριες από ολόκληρο τον κόσμο ε, παρουσία του βασιλέως ο οποίο εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τη συζήτηση που γίνεται για την κατάργηση της θανατικής ποινής με πρωτοβουλία νομικών, κοινοβουλευτικών και μελών της κοινωνίας των πολιτών. Έτσι φάνηκε ότι ορίμασε η συζήτηση για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε το κοινοβουλευτικό δίκτυο στην τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία, να ενισχύσουμε το συντονισμό στο ευρύτερο Μαγκρέπ, αλλά και στην Αφρικανική Ήπειρο, να εμβαθύνουμε τις εθνικές συζητήσεις για την κατάργηση της θανατικής ποινής υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου γιατί το Μαρόκο μετά από όλε αυτέ τι προσπάθειε και του αγώνε τη Κοινωνία των πολιτών αξίζει να κάνει αυτό το βήμα και να περάσει την κατάργηση τη θανατική ποινή. Και για πρώτη φορά έχουμε τον Υπουργό ε, δικαιοσύνη του Μαρόκου, τον κύριο Μοχάμετ Οζάρ, που είναι γνωστό ε, ακτιβιστή ε, κατά της θανατικής ποινής. Και αυτό είναι πολύ θετικό σιωνός. Η παρουσία του Υπουργού εδώ είναι ένα βήμα που μας φέρνει πιο κοντά στο στόχο μας. Να κάνουμε το Μαρόκο χώρα που θα καταργήσει τη θανατική ποινή. Περιμένουμε από εσάς, Υπουργέ, να δώσετε κάποια θαρρυντικά σημάδια προς την κοινωνία των πολιτών ότι θα υλοποιηθεί αυτός ο στόχος που είναι ένας στόχος που μας είναι ιδιαίτερα προσφυλής. Επίσης θα είναι ένας ιονός και ένα σημάδι ότι η Αφρικανική Ήπειρος θα απαλλαγεί από τη θανατική ποινή και θα δώσουμε ένα μήνυμα προς όλο τον κόσμο. Εύχομαι καλή επιτυχία στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Merci, Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που μας υπενθυμίσατε τις προεργασίες ε, και όλες τις αργότερες προσπάθειες που οδήγησαν στο σημερινό συνέδριο. Και κατά την τελετή έναρξη του Συμβουλίου ε, υπενθυμίσαμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται. Η τελετή λήξη θα γίνει το βράδυ στο ε, Μέγαρο Καλό Τεχνών, στο Μποζάρ. Βέβαια, χωρί τη δική του δέσμευση δεν θα φτάναμε εδώ σήμερα. Ο Ρομπέρ Πατεντέρα ήταν υπουργό δικαιοσύνη και το 1981 πρωτοστάτησε στον αγώνα για την κατάργηση τη θανατική ποινή στη Γαλλία. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι τότε 69% του γαλλικού πληθυσμού ήταν υπέρ τη θανατική ποινή. Θα ακούσουμε το μήνυμα του από το βίντεο. αγαπητοί μου φίλοι και σύντροφοι, λυπούμε που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας. Σήμερα κάποια απέσια μικρόβια με εμπόδισαν από το να ταξιδέψω. Αλλά δεν πειράζει. πάντοτε με ιδιαίτερη ε, ε, αλληλεγγύη προς τους έρμαχους της κατάργησης θέλω να σας απευθυνθώ στο μήνυμά μου. Σήμερα σε αυτόν τον κόσμο με τόσες δυσκολίες, τόσες εντάσεις, τόση, αγριότητα πολλές φορές είναι σαφώς ε, σωστός σκοπός η κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίω. Ήδη έχει επιτελέσει σημαντική πρόοδο σε κάποια κράτη αυτό δεν φαίνεται να φτάνει βέβαια, αλλά πρέπει εμείς ως υπέρμαχοι της κατάργησης να συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ήδη γίνει πλειοψηφία σε επίπεδο διεθνών συνόδων και συνελεύσεων. Και διαρκώς αυξάνεται ο αριθμός όσων υπερασπίζονται την ε, κατάργηση της θανατικής ποινή. Μαρτυρία σχετική, ξεκάθαρη μαρτυρία, προσφέρει το δικαιοστάσιο για την εκτέλεση της θανατικής ποινής. Με όλα τα αυτά δεν θα πρέπει να ξεχαστούμε σε κάποιο είδους ε, εφορία και ενθουσιασμό πριν ε, στην επίτευξη του στόχου μας, να υπογράψουμε όλη την ε, κατάργηση της θανατικής ποινής παγκοσμίω. Όποιος κοιτάξει προσεκτικά τα σημερινά στοιχεία και το θυμάμαι στη Γαλλία ήμουν από τους πιο ισχυρούς υπέρμαχους το 81 και περάσαμε από τις λίγες χώρες το 140, του 1981 στις 140. Ήμασταν μόλις σε 35 τότε. Πρέπει να δούμε λοιπόν τα πράγματα ξεκάθαρα, αλλά ταυτόχρονα να πούμε ότι σε μια από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου. Πολλοί ακόμη είναι υπέρμαχοι της θανατικής ποινής και υπάρχουν χώρες που την προβλέπουν τη θανατική ποινή κανονικά στο νομικό τους οπλοστάσιο. Μεγαλύτερο και χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η Κίνα. Η Κίνα που φαίνεται ότι διατηρεί ακόμη το φρικαλαίο ρεκόρ εκτέλεσης της θανατικής ποινής. Οι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα. Η Ινδία, που εμείς νομίζαμε ότι οπωσδήποτε θα ήταν η επόμενη χώρα που θα καταργούσε τη θανατική ποινή. Αλλά τη βλέπουμε να ταλαντεύεται, το ίδιο και η Ιαπωνία. Βλέπουμε επίσης ότι μεταξύ των μουσουλμάνων φίλων Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται στην, στα, πρώτη θέση των ε, απάνθρωπων ρεκόρ της εκτέλεσης θανατικής ποινής και σκέφτομαι παραδείγματα όπως το Ιράν ή η Σαουδική Αραβία που θανατώνουν τους ίδιους τους πολίτες τους. Θα μπορούσα να αναφέρω κι άλλα. Παραμένουν λοιπόν αλόβητα κάποια οχυρά, κάποιοι προμαχώνες της θανατικής ποινή. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ποιο είναι το δικό μας το καθήκον. Πρέπει να ταχθούμε ε, στο πλευρό αυτών των υπερμάχων ε, στα κράτη αυτά, ε, των υπερμάχων της κατάργησης και να τους υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο. Όπως επίσης πρέπει να ακουστεί η φωνή μας για κάθε περίπτωση, κάθε μια εκτέλεση της θανατικής ποινής ξεχωριστά. Είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Δεν θα έχουμε ε, ολοκληρώσει τον αγώνα μας εάν δεν πετύχουμε την πλήρη και παγκόσμια κατάργηση, αλλά παραμένει σίγουρα και δύσκολος ο αγώνας αυτός. Πρέπει να κινητοποιηθούμε για να, ε, κινητο... για να ε, ηγηθούμε του κινήματος των υπερμάχων και ευχαριστώ όσους ακόμα κάνουν αυτή την προσπάθεια, δίνουν αυτόν τον αγώνα και προσπαθούν να καταπολεμήσουν τη μάστιγα της θανατικής ποινή. Σε καμία στιγμή του αγώνα δεν θα ε, είναι αρκετή η προσπάθεια των υπερμάχων της κατάργηση θανατικής ποινής ε, πριν ολοκληρωθεί πλήρως ο σκοπός της παγκόσμιας κατάργησης. Εύχομαι απλώς ότι θα συνεχίσει να συγκεντρώνει περισσότερο κόσμο το κίνημά μας, να μεγαλώνει και αυτό εξαρτάται από εσά από εσά τους ίδιους που στην καθημερινή σας ε, μάχη και αγώνα αγωνίζεστε κατά της απέσιας, της φρικτής θανατικής ποινής. Είναι και παραμένει η απόλυτη άρνηση και καταπάτηση του πρώτου και ύψης του ανθρώπινου δικαιώματος, του δικαιώματος στη ζωή. Ευχαριστώ για τον αγώνα σας και να είστε βέβαιοι ότι έχετε την αμέριστη και διαρκή υποστήριξή μου. Σας λέω αντίο και εις το επανειδήν μέχρι το επόμενο συνέδριο. Ευχαριστώ. Και τώρα να απαντήσουμε σε αυτή την έκκληση δράσης ε, του Πρόεδρου Μπαρεντέρ. Έχετε αυτό το χάρτινο γάντι στα έγγραφά σας Παρακαλώ βάλτε το και σηκώστε το χέρι σας για να βγάλουμε φωτογραφία. Σηκωθείτε αν θέλετε. Παρακαλώ, σηκωθείτε. σηκωθείτε. Are you ready? Είμαστε έτοιμοι? Σχεδόν. Ωραία. Περιμένουμε να σηκωθούμε όλοι. Ποιοι είναι κατά της θανατικής ποινής. Σηκώστε το χέρι σας. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας σε αυτή την ανακτήρια εκδήλωση. Και σας υπενθυμίζω την καταπληκτική έκθεση φωτογραφιών πρώην θανατοποιητών στον πρώτο όρφο του κτηρίου. Καλείστε όλοι σε μία εκδήλωση από τις 7 το βράδυ και το πρόγραμμά μας είναι πολύ πλούσιο. Ε, Παρακαλώ, διαβάστε το από τις 3 το απόγευμα Συνεχίζεται η συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια για το ρόλο του ιδιωτικού τομέα για την κατάργηση της στρατικής ποινή. Παρακαλώ να συμμετάσχετε όλοι. Κατάργηση της ε, θανατικής είναι ένας καθημερινός αγώνας. Πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει κόσμος χωρίς θανατική ποινή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ του διοργανωτέ στην οργάνωση όλοι μαζί κατά τη θανατική ποινή, στον Παγκόσμιο Συνασπισμό κατά τη θανατική ποινή. Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που φιλοξενεί αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε το Βέλγιο. Σα ευχαριστώ που μα ακούσατε για τη συμμετοχή σα. Ευχαριστούμε και του συναδέλφου και όσου μα ε, παρακολουθούν στο ίντερνετ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνω τη συνεδρίας.